Uh, Καλημέρα σας, κυρίες ε, και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε αυτήν την διακοινοβουλευτική ε, διάσκεψη που φιλοξενεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών για την εφαρμογή του πακέτου προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με μεγάλη μου χαρά σας ε, καλωσορίζω, παρακαλώ καθίστε και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά της ε, διερμηνίας. Τα ελληνικά βγαίνουν από το κανάλι 7 για να παρακολουθήσετε την συζήτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές των κοινοβουλίων. Είναι ευχαριστησή μου ως ε, της ε, έκθεσης για τον Γενικό Κανονισμό προστασία Προσωπικών Δεδομένων να ξεκινήσω αυτήν την συζήτηση. Με χαρά σας καλωσορίζω στην πολύ σημαντική αυτή συνάντηση και χαίρομαι για το ότι έχουμε σήμερα 35 εθνικούς ε, βουλευτές ε, και γερουσιαστές από 17 χώρες και χώρες μέλη και από μια χώρα μέλος ε, της, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, την Νορβηγία. Στο θέμα μας λοιπόν, στις 27 Απριλίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό 2016 679 και την οδηγία 680 του 2016 που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων για τις διοκτικές αρχές. Έτσι πετύχαμε μια μεγάλη αλλαγή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων για να έχουμε ένα σύγχρονο και εύρωστο νομικό πλαίσιο. Το νέο αυτό πακέτο προστασίας δεδομένων ευθυγραμμίζει το πλαίσιο αυτό με την συνθήκη της Λισαβόνας και το εξυγχρονίζει για να λάβει υπόψη τις εξελίξεις ε, στην τεχνολογία και τις προκλήσεις ε, της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Είναι η ευθύ νόμη Σημαίνει ότι υπάρχει ένα νέο ενιαίο στιβαρό πλαίσιο σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης που ενισχύει τα δικαιώματα των ατόμων στην προστασία προσωπικών δεδομένων και αντικατοπτρίζει ακριβώς το ότι πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Αφενός, ο κανονισμός καθορίζει ενιαίους κανόνες για μια ενιαία εφαρμογή των κανόνων για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και έτσι οδηγούμαστε σε ίσους όρους ανταγωνισμού και ομοιόμορφη προστασία των ατόμων. Και από την άλλη, η οδηγία δημιουργεί ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων για περιπτώσεις διοκτικών αρχών στο εσωτερικό πλαίσιο αλλά και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικαθιστά τα διάφορα νομικά καθεστώτα που υπήρχαν πρώτη συνθήκη της Λισαβόνας. Για τις περιπτώσεις που δεν αφορούν τις διοκτικές αρχές ισχύει η γενική οδηγία ενώ ο κανονισμός θα ισχύει από τις 25 Μαΐου τρέχοντος η οδηγία για την αστυνομία θα ισχύει από τις 6 Μαΐου καθώς τότε εκπνέει η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν την ομοθεσία τους. Τα εθνικά κοινοβούλια είχαν εμπλακεί κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών στην έγκριση της εθνικής νομοθεσίας. Λόγω του κρίσιμου ρόλου τους στην διαδικασία αυτή, τα εθνικά κοινοβούλια βρίσκονται σε μια μοναδική θέση για να μοιραστούν μαζί μας τις θέσεις τους για το πακέτο αυτό προστασίας δεδομένων. Όμως, παρά την μεγάλη μεταβατική περίοδο που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη, είναι ενισχυτικό το ότι πολλά κράτη-μέλη δεν θα τα καταφέρουν με τις προθεσμίες του Μαΐου, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τον σεβασμό αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Η συνάντησή μας λοιπόν έχει οργανωθεί με τέσσερις συζητήσεις. Έχουμε τη θεσμική πτυχή, τον αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, την τεχνολογική καινοτομία και τέλος την εφαρμογή της αστυνομικής οδηγίας. Όλοι μας οι ομιλητές σήμερα εμπλέκονται με τα θέματα αυτά σε διαφορετικές πτυχές. Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής, ε, παρακαλώ, σημειώστε πως υπάρχει ε, διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες Ένωσης ε, πλην των Ιρλανδικών. Θα ήθελα τώρα να σας υπενθυμίσω το πώς θα γίνει η συζήτηση. Θα δίνουμε τον λόγο εναλλάξ σε δύο εθνικούς βουλευτές και σε έναν εθνικό βουλευτή και σε έναν ευρωβουλευτή μέχρι να εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών. Σας παρακαλώ λοιπόν να συμπληρώσετε τα έντυπα για να ζητήσετε τον λόγο, τα οποία σας μοιράζουν αυτή τη στιγμή και να τα δώσετε στην γραμματεία κατάλογος ε, των ομιλητών θα σχηματιστεί με αυτά τα έντυπα, με τη σειρά που έρχονται στη γραμματεία. Ε, και βεβαίω μπορείτε να μου κάνετε οι ευρωβουλευτέ ένα νόημα ω συνήθω για να ζητήσετε τον λόγο. Σημειώστε παρακαλώ ότι αναλόγως με τον αριθμό των ομιλητών ε, ίσως χρειαστεί να περιοριστεί ο χρόνος ομιλίας για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Συνήθως εδώ οι ομιλητές μιλάνε για δύο λεπτά. Τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι μετά στο μεσημεριανό διάλειμμα θα έχουμε γεύμα στον δεύτερο όροφο. Μετά από αυτές τις ε, αρχικές ε, παρατηρήσεις ε, να πω και εγώ δύο λόγια ότι πριν από τη θέση ενισχύ του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων είναι σαφές ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα προστατεύσουμε βεβαίω το θεμελιώδε μας δικαίωμα στην ιδιωτικότητα καλύτερα από ό,τι πριν, αλλά πλέον μιλάμε και για ένα παγκόσμιο πρότυπο το οποίο θα ακολουθήσουν πολλές εταιρείε παγκοσμίω και πολλές χώρες ανά τον κόσμο ήδη ακολουθούν με παρόμοιες διατάξεις ή έχουν ήδη εγκρίνει παρόμοιες ε, διατάξεις. Ε, αυτά τα λόγια λοιπόν. Να ξεκινήσουμε τώρα με το πρώτο τμήμα της ε, συζήτησής μας όσον αφορά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις θεσμικές πτυχές. Τιμή μου λοιπόν που καλωσορίζω την κυρία Ανδρέα Γέλνικ, επικεφαλής της Αυστριακής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και νεοεκλογής ε, πρόεδρο της ε, ομάδας εργασίας του άρθρου 29 δίπλα της, η κυρία Κατερίνα Ζημέλοβιτς από το Ίδρυμα Πανόπτικων ε, και αντιπρόεδρος του ΕΔΡΙ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Ψηφιακών Δικαιωμάτων και δίπλα της η κυρία Κριστίν Ενιών Αλίδα βουλευτής. Σας καλωσορίζω λοιπόν κυρίες μου και θα δώσω τον λόγο πρώτα στην κυρία Γέλινεκ για 10 λεπτά. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόσωπε, ε, κύριε πρόεδρε με συγχωρείτε. Καλημέρα σε όλες και όλους κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Δεν θα προχωρήσω σε πολλά εισαγωγικά λόγια, θα σας μεταφέρω στον κόσμο μιας μικρής αρχής προστασίας δεδομένων και στην αρχή του άρθρου 29. Όταν λέει ο πρόεδρος ότι προδιετίας τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός, αυτό είναι αληθές. Όμως οι επιχειρήσεις είχαν διετή προθεσμία για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του κανονισμού. Και όχι μόνο οι επιχειρήσει, αλλά και οι αρχές προστασίας δεδομένων. Ας αρχίσουμε με τα πιο σημαντικά που κάναμε εμεί στην Αυστρία. Κάναμε ασκήσεις χάρτου ήδη από πέρσι και δοκιμάσαμε τον One work stop ε, μηχανισμό σε συνεργασία και με άλλες προστα... αρχές προστασίας δεδομένων, δηλαδή την Ουγγρική και τη Λουξεμβουργική, και είδαμε ένα πράγμα, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάγνωση, ερμηνεία και σχολιασμό νομοθετικών διατάξεων και στην εφαρμογή του στην πράξη. Ήταν λοιπόν σημαντική η άσκηση αυτή και θα μας βοηθήσει από τις 25 Μαΐου και πλέον και πέρα να εφαρμόζουμε τους μηχανισμούς One Stop Shop τι άλλο κάναμε μέσα στα δύο αυτά χρόνια. Ενισχύσαμε, αφού αλλάξαμε πρώτα και προσαρμόσαμε τους εσωτερικούς μηχανισμούς και την εσωτερική δομή της αρχής, θα αρχίσουν να ισχύουν αυτά από τις 25 Πέμπτου. Οι συνάδελφοί μας εκπαιδεύτηκαν, που εργάζονται στην αρχή μας δηλαδή. Είχα συμμετάσχει άλλωστε στην σύνταξη του κανονισμού. Αναθέσαμε σε κάθε ένα από τους συνεργάτες μας να εξοικειωθεί με κάθε ένα από τα κεφάλαια του κανονισμού. Συντάξαμε και εσωτερικές κατευθυντήρες γραμμές, επεξεργαστήκαμε νέους διαδικαστικούς κανόνες και στο εθνικό επίπεδο, γιατί είναι πολύ σημαντικό τώρα είτε να προετοιμάζουμε την website για το 25η Πέμπτου και να προσαρμόσουμε όλα τα εθνικά έντυπα. Δηλαδή κάναμε πολλή δουλειά, όπως αντιλαμβάνεστε. Φτιάξαμε και τον λεγόμενο λευκό κατάλογο, λευκή λίστα, που έχει ολοκληρωθεί πλέον για την Αυστρία και θα περιβληθεί και αυτή τον μανδύα του κανονισμού. Δηλαδή είναι η λίστα όπου οι αρχές δεδομένων, οι εθνικές αρχές δεδομένων δηλαδή, λέγουν για ποια πράγματα δεν χρειάζεται ε, πρώτερη ανάλυση των ανακόνων προστασία δεδομένων. Και προσλαμβάνουμε και νέους συνεργάτες οι οποίοι θα αρχίσουν να εργάζονται παροιμήν από την 1η έκτου. Το Αυστριακό Κοινοβούλιο πλέον ήδη από τον Ιούλιο του 2017, 7ο του 2017 δηλαδή, ενέκρινε το σχετικό εθνικό νόμο και βεβαίως χρειάστηκε πρώτα να συνηθίσουμε και εμείς στην εφαρμογή του. Θα αρχίσει και αυτός να εφαρμόζεται από την 25η Πέμπτου και σε αυτόν βεβαίως εκπαιδεύσαμε τους συνεργάτες μας. Και βεβαίως δεν σας κρύβω ότι τα μελλοντικά μας καθήκοντα θα αναφέρονται όχι μόνο Μάλλον, θα είναι πολλά και διαφορετικά, όχι μόνο επιχειρήσεις, αλλά και εμείς. Τα λευκά πεδία που βλέπετε στον πίνακα τώρα είναι τα καθήκοντα που έχουμε ήδη. Αντιμετώπιση δηλαδή καταγγελιών, πραγματογνωμοσύνες και ατομική παροχή συμβουλών και ατομική σύνταξη εγγράφων για την εφαρμογή, για τον σεβασμό των δικαίων. Ό,τι βλέπετε τώρα γκρίζο είναι τα νέα καθήκοντα τα οποία καλούμεθα να αναλάβουμε. Δηλαδή, ως αρχή προστασία δεδομένων λαμβάνουμε και εμείς έναν αριθμό νέων καθηκόντων. Ελπίζω δε ότι είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι από τα σημαντικότερα καθήκοντα θα είναι και στην συνεργασία με άλλες αρχές προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την αρχή του One Stop Shop, της ενιαίας θηρίδας δηλαδή. Είναι ήδη σωστό ότι δεν χρειάζεται πλέον οι καταγγελίε να μεταβαίνουν από χώρα σε χώρα και από αρχή προστασία δεδομένων σε άλλη αρχή προστασία δεδομένων εντό τη Ευρώπη. Ω αρχέ προστασία δεδομένων εμεί κάνουμε το τρέξιμο. Όμω δεν είναι μόνο οι εθνικέ αρχέ που έχουν προετοιμαστεί για την θέση σε ισχύ του βασικού κανονισμού προστασίας δεδομένων. Και η ομάδα εργασίας άρθρο 29 έχει κατάλληλα προετοιμαστεί και όχι μόνο η ομάδα, αλλά ιδίω έχει φροντίσει να εκδώσει κατευθύνες γραμμές για λογαριασμό των επιχειρήσεων, 14 έως τώρα, αφενός την μελέτη δικτύπου, ε, ε, την, μετα... την δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων και ούτω καθεξής. Αυτά μπορείτε όλα και να τα αναγνώσετε, αν επιθυμείτε, στην ε, σελίδα μας στο διαδίκτυο. Και τα έχουμε και στα αγγλικά και στα γερμανικά. Βεβαίω εκεί δημοσιεύουμε και πολλά άλλα έγγραφά μας. Τι άλλο κάναμε στην ομάδα εργασίας 29, το άρθρο 29 δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια, με την σημαντική ενίσχυση του EDBS, δημιουργήσαμε και ε, προετοιμάσαμε τη γραμματεία ADPB, δηλαδή πρόκειται για τη μονάδα εκείνη η οποία θα υποστηρίξει το έργο προστασίας δεδομένων στο ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Και ως γνωρίζετε εξάλλου, το European, το European Data Protection Board είναι νέα ανεξάρτητη αρχή με αποφασιστική αρμοδιότητα. Τι άλλο κάναμε. Βεβαίως, εσωτερικά εντό τη αρχής προστασίας δεδομένων και μεταξύ αρχών προστασίας δεδομένων έχουμε προετοιμαστεί για την εφαρμογή του μηχανισμού της ενιαίας θηρίδα. και έχουμε συνεργαστεί και με εκπροσώπους μας σε ομάδες εργασίας. Αυτή η στενή συνεργασία των αρχών προστασίας δεδομένων, όπως σας εξήγησα, δεν γίνεται μονάχα σε ολομέλεια, αλλά όπως και τα προηγούμενα χρόνια περισσότερο όμως τώρα, εντονότερα τώρα, σε ομάδες εργασίας για να προετοιμάσουμε την θέση σε εφαρμογή του βασικού κανονισμού προστασίας δεδομένων. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων υποστηρίζεται από τη Γραμματεία, όπως εξήγησα πριν, και θα συνεργάζεται στενά και συνεργάστηκε συχνά με την EDPS και EDPB. Θα έχει την υποστήριξη της Γραμματείας, λοιπόν, υπό την αποκλειστική εποπτεία του Προέδρου και του Συμβουλίου. Αυτό είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του Συμβουλίου αφενός και αφετέρου βέβαια και των ανεξάρτητων αρχών προστασίας δεδομένων. Τι μπορούμε τώρα εμείς να κάνουμε στο μέλλον ως Συμβούλιο, όχι μόνο να ε, εκδίδουμε γνωμοδοτήσεις ως συμβουλευτικό όργανο όπως έως τώρα, αλλά και binding decisions, δηλαδή δεσμευτικές αποφάσεις. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα, Τήρησα τον χρόνο μου όπω θα προσέξατε κύριε Πρόεδρε και είμαι βεβαία ότι ε, τα λεπτά που εξοικονόμησα θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη συζήτηση. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Γέλνικ και πράγματι βρισκόμαστε μέσα στα χρονικά πλαίσια, οπότε θα έχουμε πράγματι την ευκαιρία να συζητήσουμε μετά. σα ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει τώρα η κυρία Σιμιέλ, Λιβίτς Για 10 λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη μου χαρά σας απευθύνω το λόγο, ιδίως για ένα θέμα που με απασχολεί τόσο πολύ, ως ε, νομομαθής και υποστηρικτρία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Χαίρομαι πολύ για την πρόοδο που έχει λάβει το θέμα και ότι γίνεται τώρα πραγματικότητα ο κανονισμός σε δύο εβδομάδες. Θέλω να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση από τη σκοπιά των πολιτών οι οποίοι υποτίθεται ότι βρίσκονται στην καρδιά του νέου κανονισμού και όχι μόνο με την ενίσχυση υφιστάμενων δικαιωμάτων αλλά και με τη δημιουργία νέων, αλλά και ιδίως με την επιβολή τους. Στο σύντομο διάστημα που έχω στη διάθεσή μου θα ήθελα να σας εξηγήσω πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση ε, της προσπάθειας αυτής, τώρα μόλις δύο εβδομάδες πριν από την θέση σε εφαρμογή. Τρία βασικά ε, σημεία. Πρώτον, εγγύησεις, safeguards, που υποτίθεται ότι θα αυξήσουν την διαφάνεια της προστασίας δεδομένων και την δεύτερον redress mechanism, δηλαδή μηχανισμούς αποζημιώσεων και τρίτον το μέλλον του κανονισμού ηλεκτρονικής e-privacy, ε, που είναι το άλλο σκέλος ε, δηλαδή. Για το πρώτο θέμα, ε, αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν ε, μεγάλες βελτιώσεις στον γενικό κανονισμό σε σύγκριση με τον προηγούμενο καθεστώς ειδικά όσον αφορά τον κατάλογο των πληροφοριών που μπορεί να δοθεί στα άτομα. Θεωρώ ότι ως άτομα θα ενημερωνόμαστε για τέτοιες πτυχές όπως ε, η πηγές των δεδομένων, οι κατηγορίες ε, των ε, δεδομένων, το προφίλ μας, όλα αυτά είναι σημαντικές ε, βελτιώσεις, ειδικά στο πλαίσιο των υπηρεσιών στο διαδίκτυο και ενός οικοσυστήματος διαφημιστικού που έχει οικοδομηθεί με τρόπο καθόλου διαφανή, όπως βλέπουμε στην περίπτωση του Facebook και σε άλλες υπάρχουν και κάποιες πολιτικές ανησυχίες αλλά τώρα οι πολίτες ε, έχουν ε, την δυνατότητα να ανακαλύψουν πώς ε, συλλέγονται οι πληροφορίες αυτές στην, στις Επίση Επίσης σημαντικό είναι ότι μπορούμε να έχουμε ένα, δεδο... ένα αντίγραφο των δεδομένων μας το οποίο μπορούμε και να μετακινήσουμε κιόλας. Σημαντικό αυτό και για τον ανταγωνισμό τούτου λεχθέντος βεβαίως βλέπω κάποιες προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των δεδομένων, όσον αφορά την διαφάνεια. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε δύσκολες νομικές μάχες για το πώς γίνεται αντιληπτή η ασφάλεια στο πλαίσιο δημιουργίας προφίλ και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν πολλές εταιρείε οι οποίες κάνουν αυτό το οποίο λέμε η δημιουργία γενικών προφίλ, χωρί να λαμβάνουν όμως αυτομάτως αποφάσεις. Δηλαδή ανακαλύπτουν ε, χαρακτηριστικά και προβλέπουν ε, συμπεριφορές χωρίς όμως να προχωρούν σε δεσμευτικές αποφάσεις. Είναι πολύ αβέβαιο εδώ πώς θα εφαρμοστούν οι διατάξεις περί διαφάνειας. Δηλαδή, εάν αρκεί για τις εταιρείε να πει κανείς ναι, σχηματίζουμε το προφίλ σας και να σταματήσουμε εκεί ή εάν θα υπάρχουν μηχανισμοί για να ζητήσουμε περισσότερες ε, πληροφορίες. Αυτή είναι η πρώτη ανησυχία την οποία ε, έχω ως δικηγόρος ε, στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι να αντιληφθούμε το σκεπτικό δημιουργίας προφίλ στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δηλαδή ακόμα και αν έχουμε κάτι που το οποίο δεν είναι παραδείγματο χάρη μια αξιολόγηση επιστολιπτική ικανότητα, αλλά αφορά τι ειδήσει που λαμβάνουμε στο Facebook. Ακόμα και αν συμφωνούμε νομικώ ότι πρέπει να αποκαλυφθεί το σκεπτικό αυτών των αποφάσεων, πώ γίνεται αυτό όταν μιλάμε για μηχανέ οι οποίε μαθαίνουν για αλγοριθμού οι οποίοι είναι πολύπλοκοι και δεν παρουσιάζονται σε ένα ε, φύλλο Excel, αλλά έχουν πολύπλοκες υπολογιστικές διαδικασίες. Αυτό θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς, για την ερμηνεία και την εφαρμογή του νέου νόμου. Όταν μιλάμε για φορητότητα των δεδομένων, το βλέπουμε αυτό ήδη στην περίπτωση του άρθρου 29. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το όριο μεταξύ δεδομένων που έδωσε το υποκείμενο τα δεδομένα τα οποία δημιουργήθηκαν από την χρήση της υπηρεσίας και δεδομένα τα οποία δημιουργήθηκαν από την εν λόγω εταιρεία. Και αυτή είναι η τρίτη κατηγορία δεδομένων που ίσως είναι η πιο προβληματική για τον ε, κόσμο και ακριβώς ε, είναι αυτό το οποίο με ανησυχεί για το πώς στην πράξη θα γίνεται αυτή η φορητότητα και μάλιστα προς όφελος των υποκειμένων δεδομένων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανακύπτουν αυτές οι προκλήσεις και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τα λύσουμε συνεργαζόμενοι για να ενισχύσουμε τα άτομα και όχι να εξασθενήσουν ε, ακόμα περισσότερο τα δικαιώματά τους. Τώρα, Μιλώντα βεβαίω για τι διαδικασίε προσφυγής και εδώ πέρα υπάρχουν κάποιε σοβαρέ ε, νίκε. όσον αφορά παραδείγματο. χάνει το πεδίο εφαρμογή του νέου νόμου. Θα υπάρχει δηλαδή ο γενικό κανονισμό ο οποίο θα ισχύει για όλε τι εταιρείε που επεξεργάζονται δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών ανεξαρτήτως του που βρίσκονται αυτές οι εταιρείε. Σημαντικό επίσης το ότι έχουμε μηχανισμούς όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να επιλέγει κάποιος ε, χώρες και ε, να ξαναζήσουμε αυτό το οποίο είχαμε με το Facebook στην Ιρλανδία, που μάλλον δεν θα είχε συμβεί σε άλλες χώρες που ερμηνεύουν διαφορετικά τον νόμο. Οπότε αυτή είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι πολίτες θα μπορούν να πάνε στα δικαστήρια απευθείας χωρίς να προσφεύγουν στις αρχές ε, προστασίας δεδομένων. Αλλά και αυτές οι διαδικασίες στην πράξη θα εξαρτηθούν από το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα είναι τα εθνικά θεσμικά όργανα. Και βεβαίω αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λύσουμε εδώ μέσα, αλλά εμείς ε, οι υπερασπιστές των πολιτών θα δούμε οπωσδήποτε αυτήν την ε, πρόκληση να ανακύπτει και βεβαίως ε, ήδη ε, δεν ξέρουμε σε ποιο φόρουμ να απευθυνθούμε, γιατί αν στην ε, Πολωνία απευθυνθούμε στον ε, επόπτη δεδομένων θα περιμένουμε δύο χρόνια. Αν πάμε στα αστικά δικαστήρια, ίσως μας παρεξηγήσουν, γιατί ο γενικός κανονισμός για τους περισσότερους δικαστές είναι κάτι το εντελώ νέο. Οπότε έχουμε προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν γρήγορα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και τα άλλα θεσμικά όργανα να παρακολουθούμε το πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν αυτά από πλευράς ερμηνείας, χρονοδιαγράμματος και τέλος για το δικαίωμα προσφυγής. Έχουμε το άρθρο 18, την παράγραφο 2, ο μηχανισμός που είχε σχεδιαστεί για μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως η δική μου για να υπερασπιζόμαστε τα ατομικά δικαιώματα. Όπως ξέρετε, τα περισσότερα κράτη-μέλη τότε δεν αποφάσισαν να εφαρμόσουν πλήρως αυτό το άρθρο και δεν δημιούργησαν διαδικασίες που θα επιτρέπουν σε κοιό να εκπροσωπούν το κοινό, το δημόσιο συμφέρον χωρίς να εκπροσωπούν κάποια συγκεκριμένα άτομα. Και από πολλές χώρες ακούω το ίδιο σχόλιο, ότι το σκεπτικό της μη εφαρμογής ε, του άρθρου 80 παράγραφος 2 ήταν κυρίως ε, να αποφευχθεί η κατάχρηση αυτού του μηχανισμού για να μην έρθουν δηλαδή πάρα πολλές ε, υποθέσεις εις βάρος εταιριών. Όμως εγώ αναμένω το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή ψηφίζουμε εφαρμογή αυτού του μηχανισμού και θα δούμε πολλές ε, περιπτώσεις κατά συγκεκριμένων εταιριών από συγκεκριμένα άτομα. Ενώ αν είχε εφαρμοστεί αυτό το άρθρο θα ήταν δυνατόν να εκδεκαστούν περιπτώσεις επί της αρχής ε, χωρίς ε, να επιτεθούμε εντό σε συγκεκριμένες εταιρείε. Ε, θα ήθελα να το τονίσω αυτό γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ε, η εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Δυστυχώς στην Πολωνία ε, δεν θα εφαρμοστεί. Τέλος, θα έχουμε μια μεγάλη πρόκληση, αυτή είναι η τελευταία μου παρατηρήση, με τον κανονισμό ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας. Ξέρετε πως υπάρχουν διάφορα ζητήματα, κυρίως λόγω του lobbying που έχει κινητοποιηθεί κατά αυτού του κανονισμού και βλέποντας το, πράγματι θα μπορούσαμε να περιμένουμε να εγκριθεί ο κανονισμός. Γιατί αν εγκριθεί ο κανονισμός τώρα υπό το, την πίεση του λόμπινγκ θα υπάρχουν κάποια παραθυράκια και εξαιρέσεις ε, για να αντιδράσουμε στις ανησυχίες ε, του κλάδου. Οπότε η ταπεινή μου συμβουλή είναι να περιμένετε λίγο πριν περάσουμε στην δεύτερη φάση. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην κυρία Κριστίν Ένιον να μας ενημερώσει για την γαλλική νομοθεσία. Έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί Ευρωπαίοι συνάδελφοι, είναι μεγάλη μου τιμή που παρεμβαίνω σήμερα για ένα θέμα τόσο σημαντικό. Σε λίγε μέρε και μετά από πολλές, ε, πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων, ο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων θα είναι ε, εφαρμοστέο και πρόκειται για μια ανεφροηγουμένου ε, νομοθεσία του θέματος. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο επηρεάζει διεθνώς. Οι τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν μια αυξημένη επαγρύπνηση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, την ελευθερία των πολιτών και την ε, ψηφιακή κυριαρχία. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνη ε, των πολιτών στην ψηφιακή, <coughs> στην ψηφιακή τεχνολογία είναι απαραίτητη. Θα περιοριστώ τώρα να σας παρουσιάσω την επιλογή των προτάσεων που έκανε η Γαλλία ε, και επίσης τα σημεία στα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε. Το, το, κείμενο αυτό είναι ένα υβριδικό κείμενο το οποίο αφήνει ε, αρκετό περιθώριο ε, εθνικού ελιγμού. Υπάρχουν λοιπόν ε, αποκλήσεις στα κρατημέλη και διάσπαση της των νομοθετικών διατάξεων και γι' αυτό τα κράτη-μέλη και οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους με αποτελεσματικό τρόπο. Το κείμενο που χτε ενέκρινε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, περιορίζει αυτό το περιθώριο λιγμών ώστε να υπάρξει όσο γίνεται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση ε, στις νομοθεσίες ε, με βάση το άρθρο 80. Ε, Μέχρι στιγμής ε, η γαλλική νομοθεσία επέτρεπε μόνο ομαδικές δράσεις, ε, ενώ η λογική ευθύνη των φορέων Σημαίνει από εδώ και στο εξής ε, ότι η, σε περίπτωση παραβίασης της ιδιωτικής ζωής των χρηστών αυτοί θα αποζημιώνονται. Πρόκειται, επίσης έχουμε από το 1978 την Εθνική Επιτροπή για την Πληροφορική και την Ελευθερία, της οποίας ε, ο τρόπος συνεργασίας με τις άλλες αρχές, ε, ευρωπαϊκές αρχές ελέγχου ορίζονται δια νόμου. Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων, ε, των ε, ερευνών, ε, καλά και των κυρώσεων θεσπίζονται και είναι εγγυημένες από την αρχή αυτή του ελέγχου. Εκεί δηλαδή όπου εμπίπτει στην αρμοδιότητα η συγκεκριμένη εταιρεία, ο υπεργολάβος για να μπορέσουν να προβούν σε ελέγχους. Το σύνολο των ε, αρμόδιων φορέων θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και καλές πρακτικές και να λαμβάνουν αποφάσεις συνενετικά εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος. Ο γαλλικός νόμος προβλέπει την προσαρμογή του εθνικού πλαισίου σε αυτά τα νέα πλαίσια ε, ε, διεθνούς συνεργασίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κοινό, κοινή ε, επιχείρηση ελέγχου στη Γαλλική Επικράτεια, τα μέλη άλλων αρχών, εθνικών αρχών, μπορούν να συνοδεύουν τους ε, εκπροσώπους της ΚΝΙΛ που προβαίνουν στους ελέγχους, το αρμόδιο δηλαδή γαλλικού <coughs> φορέα. Έτσι δημιουργείται ένα κοινό μέτωπο απέναντι σε φορείς που συχνά είναι εγκατεστημένοι εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας και έχουν επίσης σε μια αρκετά σημαντική οικονομική ισχύ ταυτότητα ε, στο άρθρο 29 θα συγκεντρώνει τους εθνικούς φορείς προστασίας αλλά και τον Ευρωπαίο Ελεγκτή Προσωπικών Δεδομένων και θα παίζει ρόλο, που θα παίζει ρόλο συντονισμού ε, και ενοποίησης της δράσης. Δύο σημεία ωστόσο θεωρώ πως ε, είναι κάπως πρέπει μάλλον να τα προσέξουμε ιδιαίτερα. Πρώτον, ο κανονισμός επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν περιθώριο λιγμού εθνικό είτε για τους ε, κατοίκους της χώρας είτε για τους υπευθύνους εκπεξεργασίας των στοιχείων. Ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία, επέλεξαν την πρώτη λύση ε, του κατοίκου, ενώ άλλες χώρες επέλεξαν την άλλη. Ε, τι θα γίνει όταν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας που είναι εγκατεστημένος σε μια χώρα που έχει επιλέξει την επιλογή των κατοίκων και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την μάλλον να εξετάσει, να ελέγξει ε, τα στοιχεία ενός ε, κατοίκου χώρας που έχει επιλέξει την άλλη επιλογή. Επίσης, ε, την ε, ηλικία, η ηλικία του ανηλίκου που μπορεί να έχει πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες. Δεν αμφιβάλλω πως ε, όλοι οι νομοθέτες έχουν επιλέξει με τον καλύτερο δυνα... τις καλύτερες δυνατές προθέσεις στην ηλικία αυτή. Ωστόσο, παραμένει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα κρατημέλη, πράγμα το οποίο θα καταστήσει περίπλοκο αυτό το μέτρο προστασίας στην εφαρμογή του. Αυτή η εφαρμογή καθίσταται ακόμα πιο περίπλοκη ανάλογα με το το αν η χώρα επικεντρώνει την προσοχή στο παιδί ή στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Θα σημειώσω τέλος ε, μία ε, πρακτική ε, λεπτομέρεια. Ο κανονισμός αυτός βασίζεται σε ένα καθεστώς ελέγχου μιας προηγούμενης αδειοδότησης από ένα προηγούμενο καθεστώς προηγούμενος αδειοδότησης σε ένα καθεστώς ε, κατάστασης υπευθύνων των ε, αρμοδίων για την επεξεργασία των στοιχείων. Και υπάρχουν ε, τελευταία πολλά αιτήματα από τους χρήστες των δικτύων να επιτρεπεί μια ανανεωμένη χρήση. Αν το σύνολο των επιχειρήσεων βλέπουν ως ευκαιρία αυτό το νέο κανονισμό, οι μικρές εταιρείε φοβούνται ότι θα είναι πολύ βαριά η εφαρμογή. Η γαλλική νομοθεσία τροποποιεί τις αποστολές και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της ΚΝΙΛ, της αρμόδιας, ε, του αρμόδιου φορέα ελέγχου. Διευρύνει δηλαδή το πεδίο αδειοδότησης αλλά και ε, του, της ε, άδειες τύπου. Επίση, οι έλεγχοι ευρύνονται και διευκρινίζονται από την νομοθεσία με δυνατότητα προσαρμογής και ενίσχυσης ε, ε, μέτρων ε, καταναγκασμού για τους ευθύνοντε οι οποίοι δεν σέβονται τις δεσμεύσει τους. Μάλιστα, οι επαγγελματικέ οργανώσεις έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα και έχουν προβλέψει τα προβλήματα που ίσως δημιουργηθούν. Προτείνονται διάφορες δράσεις για να προετοιμαστούν όσο γίνεται καλύτερα οι εταιρείε, να βοηθηθούν να μελετήσουν και να αξιολογήσουν το βαθμό συμμόρφωσης τους προς τον νέο κανονισμό, αλλά και να μπορέσουν να συνεργαστούν με αρμοδίους για την προσαρμογή και τη συμμόρφωση προς αυτό το κανονισμό. Για να καταλήξω τώρα, αυτός ο νέος κανονισμός είναι μια μεγάλη πρόοδος για την Ευρώπη όσον αφορά την ανάληψη ευθυνών των φορέων του ψηφιακού του κόσμου. Ε, τη στιγμή που ξεσπούν σκάνδαλα όπως αυτό της Cambridge Analytica και κάνουν τους πολίτες μας να ανησυχούν. Ε, ενισχύει την Ευρώπη απέναντι στους ανταγωνιστές Αμερικανούς και Κινέζους. Ε, κυρίως με λίγη ευελιξία ο κανονισμός θα μπορέσει να καταστήσει και πάλι την Ευρώπη ηγετικό, ηγετική στον παγκόσμιο ε, στην παγκόσμια τεχνολογική αρένα που φαίνεται να έχει απεριόριστες δυνατότητες. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ για αυτήν, για, για αυτές τις εισηγήσεις σας. Σας ευχαριστώ γιατί ήδη έχετε θέσει ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων που θα συζητηθούν και πριν να δώσω το λόγο στους πρώτους ε, βουλευτές θα ήθελα και πάλι να σας καλέσω να συμπληρώσετε τις ε, γαλάζιες καρτούλες αν θέλετε να πάρετε το λόγο και να τις δώσετε στη γραμματεία. τόσο οι ευρωβουλευτές όσο και οι εθνικοί βουλευτές που είστε ευπρόσδεκτοι να πάρετε το λόγο. Ο πρώτος ομιλητής θα είναι ο κύριος Κουλίτης από την Λετωνία. Σας ευχαριστώ για τις συζητήσει σας, ε, πολύ ενδιαφέρουσες και έχω να κάνω κάποιες ε, ερωτήσεις. Πρώτα στην ε, κυρία Λέχενεκ, ήταν, Χέλινεκ, συγγνώμη, ήταν εντυπωσιακά τα όσα έχετε επιτύχει, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω ποιο ήταν το τίμημα, πόσο κόστησε ολόκληρο το σύστημα για, να εγκατασταθεί. Είναι μια τοπική δημόσια υπηρεσία που έχει δημιουργηθεί. Είναι πολύ ε, κατανοητό το σύστημα, αλλά πόσο στήχησε. Ε, πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Ε, στο, προς την ε, Πολωνία εκπρόσωπο. Στη Λετωνία ε, ισχύει η προστασία από το 2000 και ο νέος κανονισμός θα το αντικαταστήσει αυτό. Ωστόσο, όταν μιλάμε για ε, προκλήσεις, <clears throat> έχουμε το Facebook, το YouTube, το, την Google, αυτές οι τεράστιες εταιρείες. Πιστεύετε προσωπικά ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κανονισμούς αντιτράστ άσχετα με το τι έχει γίνει με την υπόθεση του Facebook. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να απαντήσετε αλλά σύντομα. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Η διαδικασία δεν κοστίζει τίποτα για τον κατακέλλοντα. Η διαδικασία που ανοίγεται ενώπιον της αρχής προστασίας δεδομένων δεν κοστίζει για τον καταγγέλλοντα τίποτα. Äh, Εάν κατάλαβα σωστά την ερώτησή σας, αν εννοείται δηλαδή τώρα τι κόστισε η δόμηση της ε, αρχής, τα κάναμε εσωτερικά, χωρίς να προσλάβουμε εξωτερικούς ε, ε, συμβούλους. Δηλαδή χρησιμοποίησαμε τις γνώσεις και την εκπαίδευση των συνεργατών μας. έχω ήδη κάνει πολλές εκπαιδεύσεις σχετικά και στη βάση των συλλεκτισών εμπειριών και της συνολικής αυτής γνώσης μπορέσαμε να κάνουμε τις αναγκαίες προσαρμογές. Επομένως, δεν επιβαρύνθηκε ούτε με ένα λεπτό του ευρώ ο προπολογισμό της ε, Αυστριακής Δημοκρατίας. Για τη συγκεκριμένη ερώτηση, ε, νομίζω είναι εντάξει απάντηση, ε, θα ακούσουμε και άλλα πράγματα που σε επόμενε ερωτήσεις. Ακολουθεί ο κύριος Τράζερ από τη Σλοβενία. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω πρώτα ότι κάπως με απασχολεί αυτό που συζητούμε, διότι είναι βέβαια πολύ σημαντικό το θέμα. Αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι 25 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα αυτό, αλλά επαγγελματικά στην πολιτική δεν είμαι πολλά χρόνια. Από όσο ξέρω, στη Φιλανδία υπάρχει μια κοινοβουλευτική επιτροπή ε, που ασχολείται με το μέλλον, τη λένε του μέλλοντος. Θα έπρεπε όλα τα κοινοβούλια να τα έχουν αυτά τα πράγματα, διότι είναι κάτι που θα μα ασχολεί στο μέλλον. Αυτά τα θέματα που συζητούμε τώρα. Εγώ πολιτικός είμαι μονάχα τέσσερα χρόνια και γι' αυτό φέρνω βέβαια όμως την εμπειρία των 25 ετών. Τώρα, Facebook και οι άλλοι μεγάλοι οργανισμοί, αυτοί δεν έχουν τη βασική τους έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γνωρίζουμε αυτό όλοι. Τρίτο, ακούω συχνά να φτιάξουμε μια ευρωπαϊκή Silicon Valley. Αυτά όμως είναι ουτοπικά. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε θα πρέπει, ε, θα, θα πρέπει να είναι να φτιάξουμε τις δικές μας μηχανές αναζήτησης, ε, να αναπτύξουμε δικούς μας αλγορίθμους, όπως γίνεται στη Γαλλία, που έχουν φτιάξει μια μηχανή αναζήτησης η οποία ε, προστατεύει πολύ καλύτερα τα δικαιώματα των χρηστών, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις οδηγίες, να αρχίσουμε να συζητούμε τώρα και έστω και με 20 ετή καθυστέρηση το πώς το πώς θα θα κωδικοποιηθούν οι αλγόριθμοι στην νομοθεσία, δηλαδή πώς θα περιληφθούν στην νομοθεσία. Αυτό θα ισχύσει και για την λεγόμενη ρομποτική. Πρώτα όμως εμείς οι πολιτικοί να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι σημαίνει, ποιες ε, θα είναι οι επιπτώσεις της ε, ε, Μηχανική ευφυία. Αυτά είναι όλα ζητήματα τα οποία πρέπει να μα απασχολήσουν, απλά πρώτα να τα καταλάβουμε. Είμαστε και μια κοινωνία που γυράσκει. Άρα θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε καλύτερα του πολίτε μα ανθρώπου, για παράδειγμα, οι οποίοι δεν είναι ικανοί στην χρήση υπολογιστών. Θα πρέπει να μπορέσουν να μάθουν και αυτοί πώ να προστατεύονται. Ευχαριστώ πολύ. Thank you for your contribution. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρέμβασή σας. Να πω μόνο κάτι για αυτό το οποίο είπατε για μια επιτροπή για το μέλλον. Έχουμε και εδώ μια επιτροπή η οποία αφορά τις τεχνολογικές και επιστημονικές ε, επιλογές. Λοιπόν, να δώσω τον λόγο στην κυρία Ενιών για να απαντήσει. Ε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πραγματικά αισθάνομαι πως αυτά τα θέματα ε, είναι στην καρδιά των συζητήσεών μας και γαλλικές ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Η υπόθεση των αλγορίθμων επανέρχεται τακτικά. Έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε για να φτιάξουμε ένα σύντομο άρθρο για αυτό το θέμα, αλλά όλα όσα αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε μεταξύ μας τον συνάδελφο Βιλανή που ασχολείται με αυτό συγκεκριμένο το θέμα. Γνωρίζετε πως η Κομισιόν επίσης έχει ετοιμάσει ένα, μάλλον πρακτικά για αυτό το θέμα. Η Ευρώπη πρέπει να εστιαστεί στο μέλλον και όχι να ε, εστιάζει την προσοχή της στα όσα έχουν κάνει ήδη οι άλλοι. Πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε συλλογικά ποια θα είναι η θέση μας, ποια θέλουμε να είναι η θέση μας στο 21ο αιώνα στα θέματα αυτά που μας αφορούν και αφορούν και τις μελλοντικέ γενναίες ε, το να πούμε ότι έπρεπε να το έχουμε κάνει αυτό εδώ και 20 χρόνια, θα ήθελα να σας πω πως οι ανταγωνιστές μας δεν το έχουν κάνει ακόμα. Οπότε νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον πρέπει να αξιολογηθεί στα συν. Σας ευχαριστώ. Να απαντήσω γρήγορα για τους νόμους και τις εταιρείε ε, από τις είπα Είπα ειδικά ότι η μεγάλη νίκη του Γενικού Κανονισμού είναι ότι θα ισχύει αυτός ο νόμος για την Σιλικό και για άλλες εταιρείε. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια παρεξήγηση. Αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ο νόμος αυτός ε, θα ισχύει για οποιονδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα ανθρώπων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο Ευρωπαίων πολιτών. Το αν έπρεπε να το έχουμε κάνει αυτό πριν από χρόνια, θεωρώ ότι εμεί, εμεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ, ε, το είχαμε κάνει πριν από 20 χρόνια, γιατί οι αρχέ ε, του γενικού κανονισμού δεν είναι καινούριε. Πρόκειται για μια εξέλιξη υφιστάμενων αρχών, που δεν είναι τόσο πεπαλαιωμένε αν ε, συγκρίνεται την Γενική Αρχή με την υφιστάμενη νομοθεσία οι αρχές είναι λίγο πολύ οι ίδιες, δηλαδή ανταποκρίνονται στις ε, τεχνολογικές εξελίξεις. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, να μην δημιουργούμε ενώσεις οι οποίες θα ξεπερνιούνται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί θα βασίζονται σε πολύ συγκεκριμένη τεχνολογία, αλλά θα βασίζονται σε σωστές αρχές και για τις υπηρεσίες ε, που θέλετε να αναπτυχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε ανταγωνισμό με τις ΕΠΑ. Δυστυχώς, ευτυχώς δεν έχουμε κάποια εντολή για να αναγκάσουμε κάποιον να επιλέξει άλλες υπηρεσίες. Εάν οι αμερικανικές υπηρεσίες είναι ελκυστικές, πρέπει να ακολουθήσουμε τον κόσμο και να τους προστατεύσουμε, όχι να απαιτήσουμε ε, να δημιουργηθούν ασφαλέστερες λύσεις ε, στην ε, Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι ο κανονισμός είναι σωστή η αντίδραση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ τώρα από τους ε, σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την, το σημερινό μας πάνελ και είναι προφανές ότι το πακέτο αυτό προστασίας δεδομένων πρώτα απ' όλα Μιλάμε για ένα πακέτο που αποτελείται από δύο στοιχεία. Δεύτερον, είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδου η μετάβαση από αυτό το οποίο θα λέγαμε μια παθητική αντίδραση σε μια ενεργητική αντίδραση στην προστασία των δεδομένων. Ε, περνάμε δηλαδή σε ένα νέο καθεστώς ευθύνης για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε λοιπόν μια οριζόντια διάσταση που είναι πολύ σημαντική. Έχω όμως δύο ερωτήσεις για τους εκπροσώπους των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση των αρχών προστασίας δεδομένων. Πρώτα απ' όλα έχουμε την μετάβαση του λεγόμενου άρθρου 29 προς ένα Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Δεύτερον όμως οι αρχές, οι επόπτες δεδομένων πρέπει να είναι έτοιμοι και να ενισχυθούν στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Θα ήθελα λοιπόν να να αναφερθώ στα κράτη-μέλη. Να μάθουμε δηλαδή ποια βήματα γίνονται εν ώψη των προθεσμιών του Μαΐου έτσι ώστε οι αρχές αυτές να μπορούν να λειτουργήσουν και να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Και η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε τώρα μπροστά μας ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ολοκλήρωση του κανονισμού ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας. Γιατί τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο μπλοκάρουν αυτόν τον κανονισμό. Δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή σημαντικής νομοθεσίας που έχει μπλοκάρει το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη δηλαδή. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή εδώ των εθνικών βουλευτών για να γίνει και αυτή η δουλειά και να ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όχι μόνο να τεθεί ενισχύ, δηλαδή, αλλά να ολοκληρωθεί η εικόνα με το να υπάρχει προστασία της ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας των πολιτών στην ε, ενιαία αγορά. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Πουτλόφσκι από την Πολωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ που ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα προστασίας δεδομένων. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε η κυρία Σιμιολέβιτς και έχω κάποια σχόλια για τα οποία θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των συναδέλφων θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε έναν από τους σημαντικότερους κανονισμούς στον τομέα της προστασίας δεδομένων. Δεν ξέρω τι γίνεται στις χώρες σας, αλλά στη χώρα μου είναι κάπως άργα όσον αφορά την αντίληψη των εταιριών, όπως είπε και ο συνάδελφος από την ε, Σλοβενία, ο κ. Στρότσεκ. Ε, έτσι και εγώ δεν είμαι πολιτικός ε, εδώ και πολύ καιρό και πρέπει να σας πω ότι από τη Σκοπιά του επιχειρηματία, του ιδιοκτήτη εταιρεία. Πέρα από τις τεράστιες εταιρείε που προφανώς έχουν τους πόρους να τα κάνουν αυτά, οι μικρές εταιρείε δεν έχουν αντιληφθεί ε, το τι εστί η εφαρμογή αυτού του κανονισμού και αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ε, ότι θα πρέπει να μπορέσουν να αποφύγουν τι συνέπειε ε, μια νομική διαμάχη. Και αναρχέμαι. Αυτό γίνεται εξαιτία του ή εξαιτία τη διαδικασία που, με την οποία προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Η οποία δουλειά μας είναι η καλύτερη προστασία των πολιτών και βεβαίως να αντιληφθούν καλύτερα τα δεδομένα εταιρείε. Τι κάνουμε λοιπόν. Υπάρχει μια τεράστια δυνητική τιμωρία των εταιριών και μετά απαιτούμε αλλαγές. Ε, θεωρώ ότι δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Αντί λοιπόν να νομοθετούμε μόνο, να προτείνουμε και μία πορεία πώς θα θέλαμε να γίνει η εφαρμογή και τι θα μετρήσουμε. Εάν γνωρίζουμε ότι σε δύο χρόνια θα ισχύει ο κανονισμός και ο κόσμος θα γνωρίζει το τι σημαίνει αυτό, να πούμε ότι θα υπάρχει ένα μέτρο κατανόησης πόσες εταιρείε έχουν αντιληφθεί το τι σημαίνει αυτό. Σε ένα χρόνο να γνωρίζουμε το αν έχει γίνει αντιληπτό στι χωρε γιατί στι περισσοτερε χωρε δεν έχει γίνει αντιληπτό. Αυτό πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου, γιατί είμαστε πίσω. Και δεν μιλάω νομίζω μόνο για τη χώρα μου, στα περισσότερα μέρη τη Ευρώπη είμαστε πίσω. Όχι τόσο στην νομική πτυχή, γιατί αυτό εύκολα γίνεται από τα κοινοβούλια, αλλά στην πραγματική εφαρμογή να αντιληφθούν οι εταιρείε το τι σημαίνει αυτό, να προετοιμάσουν τι διαδικασίε στο εσωτερικό των εταιριών για τα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, καλοδεχόμενη αυτή η παρέμβαση όλοι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της καλύτερης αντίληψης των όσων γίνονται εδώ. Οπότε νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτή για να συμβεί κάτι τέτοιο. Η κυρία Κοσμοβολή από την Ελλάδα. you have to use the microphone. You can switch it on uh, on your uh, on the other side. Okay. να πατήσετε το μικρόφωνο, το κουμπάκι του μικρόφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να συγχαρώ και να επενέσω τους διοργανωτές που κάνουν αυτή τη συζήτηση ενώψη του, ε, της εφαρμογής του κανονισμού ε, στα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Ε, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις κατέστησαν αναγκαία την αντικατάσταση του ισχύοντος από το 1995 νομικού πλαισίου για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. Να θυμίσω τότε που το διαδίκτυο ε, ήταν ελάχιστα διαδεδομένο. Και αυτό το, το νομικό πλαίσιο που υπήρχε αντικαθίσταται από ένα κανονισμό συνεκτικό, ενιαίο και ε, για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης που θα, που θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και επειδή η τεχνολογία τρέχει με λιγιότητα ταχύτητα, πρέπει ομοίως να προχωρήσουμε με ταχύς ρυθμούς, θεωρώ ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει. Τώρα στη χώρα μου, στην Ελλάδα, το σχέδιο νόμου που θα ενσωματώσει την οδηγία 216-680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 στο εθνικό μας δίκαιο ε, περιέχει ε, και ο νόμος αυτός που περιέχει τα μέτρα εφαρμογής και υλοποίηση του κανονισμού είναι έτοιμος και εντός των επόμενων ημερών θα έρθει προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο. Ε, έχει προετοιμαστεί κατά τέτοιο τρόπο που να διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού. Σε αυτό το θέμα βρισκόμαστε σε καλό σημείο. Όμως, η εποπτεύουσα αρχή της εφαρμογής του κανονισμού που στην Ελλάδα είναι η ανεξάρτητη αρχή προσωπικών δεδομένων έχει ήδη μεγάλο όγκο αρμοδιοτήτων και χρειάζεται ενίσχυση οικονομική, ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων και ενίσχυση, ε, και ε, ενίσχυση των δομών για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Επίσης πρέπει να ενημερωθούν και τα δικαστήρια. Η δικαστική εξουσία γνωρίζουμε είναι μια ανεξάρτητη εξουσία και με αυτή την έννοια δεν ε, μπορεί κάποιο να παρέμβει. Είναι απαραίτητο όμω να εκπονηθούν ειδικά σεμινάρια ενημέρωση των δικαστικών αρχών. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρέμβασή σας. Βλέπω ότι έρχονται σιγά σιγά τα έντυπα για την ε, ε, λήψη του λόγου. Παρακαλείστε να συνεχίσετε εφόσον επιθυμείτε. Κύριος Δίας Τεμέρα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και ειδικά τους συμπατριώτες μου από το Γενικό Δικαστήριο και τους ε, συμβούλους που τους ε, ε, συνοδεύουν. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή ανταλλαγή απόψεων, γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να σας δώσω κάποιες εξηγήσει και ενημέρωση για τους εκπροσώπους της, της, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι στη διάρκεια της συζήτησης των διαπραγματεύσεων για την οδηγία και τον κανονισμό, το Ευρωκοινοβούλου στο πλέον του, ε, της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας ε, ε, ακολούθησε τι συνέβαινε ε, σε τομέα αυτών. Εγώ θα αναφερθώ στο τομέα εργασία στον οποίο πρωταγωνίστησα και είμαι αρμόδιος, δηλαδή επεξεργασία των στοιχείων στον ποινικό και αστυνομικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, όπως ήδη γνωρίζει ο Πρόεδρος, τα ευφυή σύνορα, Frontex, ε, είσοδος και έξοδος, Europol, Eurojust, ε, εισαγγελία, έχουμε προχωρήσει σε τέτοιο σημείο ώστε τελικά ε, χρειάστηκε να μπορέσουμε να συζητήσουμε στο μέλλον ε, τι θα γίνει αν υπάρξει κάποια παράβαση του κανονισμού και είμαστε σε θέση να προτείνουμε τροπολογίες για να προσαρμόσουμε συγκεκριμένα, ε, σε, συγκεκριμένα στις καταστάσεις που θα συναντήσουμε. Έχω, επίσης την απορία ότι σε αυτά εδώ ε, τα πάνελ που με τόση προσοχή και ε, προετοιμάσατε δεν είναι ο κύριος Μπουταρέλη σε κανένα από αυτά τα πάνελ που είναι ο αρμόδιος για την προστασία των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έπρεπε και εκείνον να τον ακούσουμε και να συζητήσουμε μαζί του κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ. Ρωτήσατε γιατί δεν είναι εδώ η EDPS, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασίας των Στοιχείων. Θέλαμε να έχουμε τις εθνικές αρχές περισσότερο σήμερα εδώ. Ε, επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Φουγκέ από το Βέλγιο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να θέσω μια ερώτηση που ανέφερε και η κυρία Ενιό το μικρόφωνο σας ε, πρέπει να ανάψετε. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να ε, επιστρέψω στα όσα είπε η κυρία Ενιού για την προστασία των ανηλίκων και να έχουμε και τη γνώμη μιας ΜΚΟ που προστατεύει τους πολίτες για αυτή την πτυχή. Ξέρουμε πώς έχουμε αφήσει ένα περιθώριο ελιγμών στα κράτη. Μπορεί να είναι εντάξει στο επίπεδο ε, σε κατάρτισης όμως τι γίνεται για να προστατευθούν οι ανήλικοι και ποια είναι η άποψη της ΜΚΟ που εκπροσωπεί ε, την προστασία των πολιτών. Θα θέλατε να απαντήσετε αμέσως. Uh, thank you for the question. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, δεν προσδίδουμε τόσο μεγάλη σημασία στο κατόφλι της ηλικία που έχει συζητηθεί τόσο έντονα, αν θα είναι 13 ή τα 13 τα 14 χρόνια. Πάντως, πιστεύω πως δεν θα προστατέψουμε τα παιδιά που πηγαίνουν online και έχουν και τις υπηρεσίες. Όσο ψηλότερο είναι το κατόφλι, τόσο, και όσο καλύτερο είναι οι μηχανισμοί για τη διαφάνεια για τον έλεγχο των χρηστών αλλά και για την εκπαίδευση των χρηστών. Ορισμένους τους έχουμε τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες να καταλήξουμε σε καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τους ανηλίκους. Δεν νομίζω πως μπορούμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους νέους με συγκεκριμένα μηχανισμούς, ακριβώς επειδή είναι πολύ δύσκολο να αποδειχτεί και να επιβληθεί η υποχρέωση της επαλήθευσης της ηλικία. Όμως, όσο πιο καλά εφαρμοστούν όλοι αυτοί οι κανόνες, τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα για τους ανηλίκους. Ah, wanted to speak also on this. Η κυρία Ενιό. Ναι. Έγινε μακρά συζήτηση στο πλαίσιο του Γαλλικού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο το ηλικίας. Εγώ ίδια είχα προτείνει τα 13 έτη, ε, προτείνοντας ότι η παιδεία πρέπει να επιβληθεί να υπερισχύσει. Τελικά καταλήξαμε στην 15 ε, έτη, αλλά επιμείναμε για ενισχυμένη κατάρτιση και ε, για το γεγονός ότι πρέπει να εκπαιδεύονται τα παιδιά από το σχολείο και από την ε, μικρότερη ηλικία στους κινδύνους της χρήσης. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με το Υπουργείο Παιδείας και τα διάφορα αρμόδια άλλα Υπουργεία Και εδώ ίσως ε, να εγκαλώ κάπως την ε, γειτόνισά μου. Λέτε πως η ε, ηλικία δεν είναι σημαντική, αλλά νομικώς πρέπει να υπάρχει μια ηλικία και άρα να υπάρχουν και συνέπειες για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν τέτοιες διαδικασίες ή όχι. Ε, μάλιστα, ευχαριστώ. Ο κύριος Ράλλο από την Ισπανία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα συνεχίσω με το θέμα που συζητάμε την ηλικία δηλαδή των ενηλίκων ε, αλλά από κάποια γενικότερη οπτική γωνία. Εμένα ένα θέμα που με ανησυχεί σε μια τέτοια αυτή την κατάσταση που είναι πραγματικά μια επανάσταση στους τελευταίους μήνες για την προστασία των στοιχείων είναι το θέμα ότι αρχίζει να φαίνεται μια κάποια απόσταση ανάμεσα στον κανόνα και την πραγματικότητα. Ο κανόνας ε, πνέεται από μια φιλοσοφία συνδυασμού μεταξύ μιας ε, ε, στρατηγικής αντίδρασης και μιας στρατηγικής πρόληψης. Αυτή η πρόληψη είναι ακριβώς ο μέγας στόχος που έχει αναλάβει αυτός ο κανονισμός ως σπουδαία καινοτομία και τοποθετούμε πολλές ελπίδες στη λειτουργία αυτού του κανονισμού, όμως φαίνεται να υπάρχουν κάποια κενά που αποδεικνύουν ότι αυτή η δραστήρια στρατηγική, η προληπτική στρατηγική θα είναι τελικά ίσως λιγότερο αποτελεσματική από ότι η πολιτική, η στρατηγική μάλλον αντίδρασης. Το είπε η Γαλλίδα εκπρόσωπος και μάλιστα το επανέλαβε μόλις ότι ο κανονισμός δεν έχει αποφύγει ένα κάποιο βαθμό που αρχίζει να φαίνεται δεν έχει αποφύγει αρκετά μεγάλο βαθμό α, απόκλησης ανάμεσα στους εθνικούς, ε, ε, ε, στις εθνικές νομοθεσίες και ιδιαίτερα όσον αφορά τους ανηλίκους. Έχουμε από 13 μέχρι τα 16 χρόνια τις Έχουμε διάφορους που έχουν αποφασίσει από την ηλικία των 13 μέχρι και των 16 ε, θεωρούν. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα όταν θα πρέπει να εγγυηθούμε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτού του κανονισμού. Και μάλιστα τα τελευταία, στις τελευταίες μέρες υπάρχει κάτι ακόμα που είναι σαφές, ότι δόθηκε, που μάλιστα το έκανε η WhatsApp. Η WhatsApp στέλνει μηνύματα στους χρήστες της που του ζητά να επιβεβαιώσουν ότι ε, συγκατατίθενται στη χρήση της υπηρεσίας αυτής και να αναγνωρίζουν μάλιστα και να δέχονται, ε, να επιβεβαιώνουν ότι, έχουν, ε, ότι είναι άνω των 16 ετών. Η άρα ευθυγραμμίστηκε με το ανώτατο δυνατό όριο και άρα θεωρεί ότι έτσι διαφεύγει του προβλήματος. Οι μικρότεροι των 16 ετών, 14, 15, 10, 12, 9 ετών που πατάνε το κουμπάκι ναι, ότι δηλαδή δέχονται αυτή την, ε, την, την, τη συγκατάθεση και ότι είναι πάνω από τα 16 χρόνια, δεν μπορεί να τους ελέγξει κανείς. Άρα λοιπόν οι εταιρείε θα πρέπει να υιοθετήσουν ε, κάποια λογικά μέτρα για να επαληθεύουν αυτή την ηλικία όταν ζητούν αυτή τη συγκατάθεση. Αυτό είναι πολύ σοβαρό στόχο για να μην δημιουργηθεί δυσπιστία ανάμεσα στου χρήστε και τον κανονισμό που τώρα αρχίζει να ισχύει και όπου ήδη διαφαίνονται τέτοιου είδους ελλείψεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα θέλατε να απαντήσετε κάποια από τις τρεις κυρίες. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας και ιδίως για την συγκατάθεση που είναι σημαντική υπόθεση να δούμε όλοι πώς κάνουν το παιχνίδι των updates στην ε, πολιτική τους οι μεγάλες εταιρείες σε αυτές τις εβδομάδες πριν αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός. Δηλαδή βάζει κανείς το σταυρουλάκι στο κουτάκι, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τίποτα όταν λέει ναι είμαι πάνω από 16 ετών. Όμως έχει διαφορά αν είσαι 10 χρόνων ή 16 ή παραπάνω. Αλλά δεν έχουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να προστατεύσουμε τους ανηλίκους όταν πηγαίνουν online. Υπάρχουν άλλοι τρόποι από την απαγόρευση. Και βέβαια δεν μπορούν να αναλάβουν ευθύνε από συμβάσεις. Η απαγόρευση όμως στην πράξη δεν πρόκειται ε, να λειτουργήσει και σε αυτά τα pop-up των διαφόρων εταιριών Πολλέ από αυτέ προσφέρουν τώρα στου πολίτε εναλλακτική συγκατάθεση. Μπορείτε τώρα ή μπορείτε αργότερα. Δηλαδή μπορείτε να προχωρήσετε και χωρίς να δώσετε συγκατάθεση. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι μια πίεση που ασκεί στον χρήστη για να δώσει τη συγκατάθεση και να νομοποιήσει κάποιες ε, πρακτικές πριν να γίνει απόλυτα εφαρμόσιμος ο κανονισμός που θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε λίγες εβδομάδες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί νομικά αυτή η πρακτική, αλλά τουλάχιστον πολιτικά θα έπρεπε να μπει κάποιο φρένο. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα έχω τέσσερις ακόμη ευρωβουλευτές, Ζίπελ, Γκόμες, Στίβενς και Ιντφέλτ. Και θα τους δώσω τον λόγο, όμως στο μεταξύ, εάν υπάρχει άλλος βουλευτής από Εθνικό Κοινοβουλίο που επιθυμεί να λάβει το λόγο, παρακαλώ να συμπληρώσει το γαλάζιο έντυπο και να το δώσει στη γραμματεία. Θα ακολουθήσει λοιπόν η κυρία Ζίπελ από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Θα ήθελα να στρέψουμε τα βλέμματα προς τα πίσω, διότι εγκρίναμε τον κανονισμό το 2016, άρα υπήρχε μια διετία για να μπορέσουν να προετοιμαστούν κυβερνήσεις, κρατικές αρχές, ε, μη κρατικές οργανώσεις και επιχειρήσεις. Η εντύπωση μου όμως είναι ότι μόλις τις τελευταίες εβδομάδες αρχίζουν κάποιοι από τους ενδιαφερομένους να προετοιμάζονται. Δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά πώς είναι δυνατόν τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες να λαμβάνει το γραφείο μου πάρα πολλές, πάρα πολύ ακριβώς διατυπωμένες ερωτήσεις, τις οποίες δεν λάβαμε ποτέ πριν. Είχαμε λοιπόν δύο χρόνια προετοιμασίας και ένας από τους στόχους ήταν να εναρμονιστούν τα πρότυπα, διότι προστασία δεδομένων υπήρχε και πριν από τον κανονισμό, αλλά ένας από τους στόχους τώρα ήταν να υπάρξει ένα ενίο πρότυπο σε όλη την Ευρώπη, ώστε να διευκολυνθούν ιδίω οι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Αλλά βεβαίω και οι πολίτε όταν, μεταβε... όταν διαβαίνουν τα σύνορα από τη μια χώρα στην άλλη. Ποια είναι η εμπειρία σα λοιπόν, για παράδειγμα, στην ομάδα εργασία σε ό,τι αφορά τις προετοιμασίες των ίδιων των χωρών μελών, για τις οποίες, για ορισμένες από τις οποίες μάλλον, ο κανονισμός μπορεί να είναι κάτι το νέο. Έχω και ένα ανακοινωθέν τύπου εδώ μπροστά μου που λέει ότι από 24 αρχές προστασίας δεδομένων που απάντησαν σχετικά με τις ερωτήσεις αυτές, μόνο 17 θεωρούν ότι είναι πλήρως εξοπλισμένες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ε, νέες προκλήσεις και ευκαιρίες του κανονισμού. Θεωρείτε ότι οι Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων είναι σε θέση να προστατεύσουν και να ε, διευκολύνουν τις επιχειρήσεις, τους χρήστες κλπ. Και μια συγκεκριμένη ερώτηση που δεν λέγεται ακριβώς στο GDPR. Τι γίνεται όμως με τις εικόνες, φωτογραφίες. Είναι μια από τις ερωτήσεις τις οποίες λαμβάνω διαρκώς. Αν πάρω μια φωτογραφία ανθρώπων που βρίσκονται στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, στο δρόμο, σε ένα κατάστημα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία, μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία για να αποκομίσω κέρδο. Και τι γίνεται με όλα τα πρόσωπα που είναι μέσα στη φωτογραφία. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα προστασία. Πώ ρυθμίζεται στι χώρε σα το ζήτημα αυτό ή παραμένει ακόμη ανοιχτό στι χώρε σα. Αυτό θα ήθελα να ερωτήσω. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Παρακαλώ αν θέλετε να απαντήσετε. Ίσως κυρία Γέλνικ πρώτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας και ιδίω ό,τι αφορά το σκέλος της ε, προετοιμασίας. Δεν βομβαρδίζετε μόνο εσείς, βομβαρδιζόμαστε και εμείς και μάλιστα ήδη τα τελευταία δύο χρόνια από τέτοιες ερωτήσεις. Βέβαια, έχει ενταθεί πολύ αυτό τις τελευταίες εβδομάδες. Όντως είναι εκπληκτικό ή τέλος πάντων κάπω ευνηδιαστικό γιατί έχουν ορισμένοι την εντύπωση ότι η τελος παντων καπω ευνηδιαστικο γιατι εχουν ορισμενη δεδομένων τους έπεσε από τον ουρανό στο κεφάλι ενώ θα πρέπει να είναι γνωστό. Εδώ και 40 χρόνια έχουμε στην Αυστρία τουλάχιστον νόμο περί προστασίας δεδομένων. Τώρα ο κανονισμός αποτελεί μία, μάλλον ένα παραπέρα βήμα μετά από την οδηγία. Θα πρέπει βέβαια σε όλες τις χώρες μέλη να προσαρμοστούν τα σχετικά πρότυπα, ώστε να μην οδηγεί το κόσμο σε αυτό που λέγεται forum shopping, δηλαδή άγρα ε, του πιο ευνοϊκού ας πούμε ε, τόπου όπου μπορεί να υπάρχει ρύθμιση. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις, ως γνωρίζουν άλλωστε εδώ και δεκαετίες, να έχουν μια ιδέα για το τι θα κάνουν και βεβαίως και ποια πράγματα θα αλλάξουν, ποιες είναι οι πρόσθετες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και ούτω καθεξής. Και καμιά φορά εμείς λέμε, κοιτάξτε, καθίστε να διαβάσετε τα κείμενα. Ο κανονισμός είναι γνωστός εδώ και δύο χρόνια. Υπήρξε μια περίοδος χάριτος, όπως ε, ζητείτε συχνά και όπως δίνετε συχνά, δύο ετών. Άρα δεν υπάρχει τίποτα το νέο. Και 25η Μαΐου δεν είναι καμία μυστική ημερομηνία, είναι γνωστή. Άλλωστε και το κείμενο του κανονισμού είναι γνωστό. Και υπάρχει και μάλιστα υπάρχει και σχολιασμό σε πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ γλώσσε. Βεβαίω ορισμένα πράγματα χρειαστεί να ξεκαθαριστούν δικαστικά, δηλαδή από το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Αυτό συμβαίνει όμως και με κάθε νομική ρύθμιση. Αυτά σχετικά με την προπαρασκευή, με την προετοιμασία. Το ερώτημα τώρα σχετικά με τις 24 αρχές προστασίας δεδομένων από τις οποίες μόνο οι 17 θεωρούν ότι έχουν επαρκή προετοιμασία και εξοπλισμό. Βεβαίω δεν γνωρίζουμε πόσες διαμεθοριακές υποθέσεις θα μας έλθουν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και χρόνια. Υπάρχει μια βεβαιότητα. Αυτό καθιστά δυνατόν το ενδεχόμενο κάποιε ε, αρχέ προστασία δεδομένων αποδειχτεί ότι δεν είναι επαρκώ εξοπλισμένε. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Ούτε και εγώ έχω καμιά κρυστάλλινη σφαίρα για να δω το μέλλον. Δεν μπορώ να είμαι βεβαία ότι και η Αυστριακή Αρχή Προστασία Δεδομένων είναι επαρκώ εξοπλισμένη. Έχουμε ζητήσει περισσότερε ε, θέσει προσωπικού από όσε λάβαμε τελικά. Αυτό βέβαια θα έχει γίνει και σε άλλες ε, χώρες μέλη, κάτι το οποίο δεν με ικανοποιεί, αλλά οφείλω να το λάβω υπόψη. Θα, κάνω κάθε, θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κανονισμού. Πέραν αυτού υπάρχει και η δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 4, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλλει σε μια υποστήριξη των αρχών προσθέσεων δεδομένων εφόσον δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Τώρα, αυτά ως συνολικότερη εικόνα. Πάντως, νομίζω, ή μάλλον να το πω ως εξής, καταρκούνται ορισμένες υποχρεώσεις δικές μας και προσθέτεται κάποιες άλλες. Σχετικά, για παράδειγμα, με μια περιφερειακή αρμοδιότητα που είχαμε και η οποία δεν είχε ληφθεί, δεν είχε δηλαδή, δεν τη είχαμε χρησιμοποιήσει επαρκώς έχουμε τώρα για τα νέα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει μια νέα, ένα νέο τμήμα. Δεν ξέρω τι είδους επιβάρυνση θα έχει αυτό το νέο τμήμα μετά την 25η Πέμπτου. ομως θεωρώ ότι είμαστε επαρκως προετοιμασμένες. Βεβαίω, αν αποδειχτεί ότι όχι, θα κάνουμε κάποια βελτίωση. Και οι χώρες μέλη έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προετοιμάσουν καλύτερα τις, ε, και να αξιοποιήσουν καλύτερα τις αρχές προστασίας δεδομένων. Και θα χρειαστούν ενδεχομένως, θα χρειαστεί ενδεχομένως τα κοινοβούλια να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις, να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν καλύτερα τις αρχές προστασίας δεδομένων. Ευχαριστώ. Η κυρία Ένιον. Η ερώτησή σας ε, περιέχει πολλά σκέλη. Όσον αφορά τις εθνικές αρχές, όπως είπα, η ΚΝΙΛ υπάρχει από το 1978. Πρόκειται για μια αρχή που ε, σιγά σιγά εξελίχθηκε και πλούτησε στη διάρκεια των ετών με νέα τεχνικά μέσα, νομικά μέσα και διάφορους εμπειρογνώμονες που ε, κάνουν, κάνει μάλιστα και δικά της ε, πειράματα. Βέβαια μετά το νέο αυτό κείμενο το φάσμα των αποστολών διευρύνεται και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Κνήλη θα χρειαστεί επιπλέον με πόρους Όλοι, όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου το έχουν συνειδητοποιήσει. Θα πρέπει να το δούμε όμως μέσα σε ένα πλαίσιο ε, δημοσιονομικό. Θα πιέσουμε ώστε οι αρχές να ε, συνεχίσουν να ενισχύουν, να ενισχύονται μάλλον στα επόμενα χρόνια έχει προετοιμαστεί εδώ και δύο χρόνια ε, ε, φτιάχνοντας ε, οδηγούς, βίντεο, οργανώνοντας διασκέψεις και προσπαθώντας να συνδεθεί με την κοινωνία των πολιτών που Έχουμε πολλά επαγγελματικά συνδικάτα ε, που ασχολήθηκαν με το θέμα για να ε, μπορέσουν να καταρτήσουν τα μέλη τους. Και εμείς στο Γαλλικό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να ε, προωθήσουμε αυτό το κείμενο στις εταιρείε και το επίπεδο προετοιμασίας βέβαια διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της εταιρεία. Όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι, οι μικρότερες εταιρείε κάποιες φορές ανησυχούν, αλλά και η αρχή αυτή έχει μέγα ρόλο συνοδευτικό. Ανέκαθεν το έκανε και θα συνεχίσει να το κάνει. Δεν θέλουμε να είμαστε τόσο ε, άκαμπτοι, αλλά βεβαίως ε, θα έχουμε μια ενισχυμένη παρακολούθηση και ε, συνοδεία. Να κάνω μια παρατήρηση. Αυτή η συζήτηση βεβαίως αφορά και την ελευθερία τις φωτογραφίες έχουμε το άρθρο 85 και την ελευθερία έκφρασης. Υπάρχει ανάγκη ε, τα κρατη να κάνουν και αυτά τη δουλειά τους με τη σειρά τους. Παρακαλώ. Ναι. Στη Γαλλία έχουμε επίσης κείμενα για το δικαίωμα στην εικόνα που αφορούν αυτήν την πτυχή και βεβαίως θα πρέπει να ζητούμε άδειε ε, για τα παιδιά. Φυσικά ε, θα πρέπει αυτό να γίνεται ακόμα και αν είναι κείμενο το οποίο είναι διαφορετικό από αυτόν τον κανονισμό, ή προϋπήρχε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε δύο ακόμα μέλη από τα Εθνικά Κοινοβούλια και μετά θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Επόμενος ομιλητής, κ. Έσκεντ από τη Γερμανία. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε τον κανονισμό αυτό και την εφαρμογή του. Όλοι βεβαίως αναμένουμε να δούμε πώς ε, θα είναι τελικά η εφαρμογή των διαφόρων θεμελιωδών αυτών δικαιωμάτων. Ένα ενδιαφέρον μήνυμα από τη Γερμανία είναι ότι σήμερα είχαμε μια καταγραφή μια κάμερα παρμπρίζ αυτοκινήτου την οποία επέτρεψε το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο ως αποδεικτικό μέσο σε δικαστήριο, πότε αν κυκλοφορώ και καταγράφω την κίνησή μου για να μπορώ σε δυνατότητα, σε πιθανότητα ατυχήματος να αποδείξω αυτό το οποίο συμβαίνει, υπάρχει η πιθανότητα πράγματι να κατηγορηθώ ότι παραβιάζω προσωπικά δεδομένα. Πράγματι στη Γερμανία όπως και σε άλλα κράτη-μέλη υπάρχει κάποια ανησυχία μετά από τα δύο χρόνια που είχαμε στη διάθεσή μας για να εφαρμόσουμε τον ε, κανονισμό. Ανησυχία για το πόσο γρήγορα τώρα θα αρχίσουν να επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές ε, πρόστιμα και προειδοποιήσεις ε, τις οποίες αποστέλουν, ξέρετε ότι έχουμε ε, μια ιδιαίτερη έφεση σε αυτό στην ε, Γερμανία και είναι κάτι το οποίο απασχολεί την ε, κοινωνία των πολιτών και τις διάφορες ενώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατόπιν ο κύριος Μαρτίν Τούλενταν από την Ισπανία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι πρόκειται για κανονισμό, για ένα θέμα το οποίο είναι ζωντανό και που εξελίσσεται διαρκώς. από μια ρύθμιση για την προστασία δεδομένων που είχαμε όλες τις χώρες μας, που ήταν ε, παρκής ίσως, αλλά δεν ήταν ομοιογενή σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια μεγάλη όθηση που βέβαια δεν θα είναι η τελευταία, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε. Εγώ ήθελα να κάνω μια σειρά παρατηρήσεων ως ε, εκπρόσωπος των βουλευτών ε, της Ισπανίας και ο κύριος Δίας Δημέρα ε, εξέφρασε ένα προβληματισμό, γιατί μιλάμε πολύ για την οδηγία, όμως για τον κανονισμό, συγγνώμη. Έχουμε όμως και την 680 και την 681 για τα θέματα προστασίας των δεδομένων των ε, ερευνών μέσω των ευρωπαϊκών οργανισμών, των ποινικών. Και είναι νομίζω σημαντικό να σκεφτούμε Ε, αν υπάρχουν απαιτήσει για την προστασία των δεδομένων που επιβάλλονται στις ιδιωτικές εταιρείε του τομέα που λειτουργούν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών αλλά και του οικονομικού κέρδους και πρέπει πολύ σαφώς να ορίσουμε τι είναι το δημόσιο συμφέρον που, των εταιριών που πρέπει επίσης να, των δημόσιων μάλλον οργανισμών που πρέπει επίσης να χειρίζονται στοιχεία αλλά με μια νομική προστασία για να αποφευθούν ε, οι παραβιάσεις αλλά και τα δικήματα κυρίως κατά των ε, ανηλίκων. Υπάρχουν ε, και διατάξεις που απαγορεύουν ε, την υπογραφή συμβάσεων από ανηλίκους. Ορισμένα, ορισμένες δε συμβάσεις που γίνονται διαδικτυακά σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, εκεί οι ενήλικοι θα πρέπει να προστατευτούν όλους ιδιαίτερως, γιατί αυτές οι συμβάσεις που υπογράφουν και που αρχίζουν να ισχύουν με βάση εθνική, την εθνική μας νομοθεσία είναι ε, άκυρες. ευχαριστώ πάρα πολύ, Γκόμες ε, από τους Σοσιαλδημοκράτες Ευρωβουλευτής. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι στον Λετωνό συνάδελφο που ρώτησε πριν ε, μήπως πρέπει να σκεφτούμε κάποια νομοθεσία για νομοθεσία περί μονοπωλίου για να καταπολεμήσουμε την δεσπόζουσα θέση κάποιων πλατφορμών όπως το Facebook, Google κτλ. Συμφωνώ απολύτως. Πραγματικά αυτό χρειαζόμαστε και περισσότερα ακόμα. Χρειάζεται φορολογία. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, όχι μόνο για να σταματήσει η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεις αλλά να υπάρχουν και ίσοι όροι ανταγωνισμού με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό εμείς οι νομοθέτες να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε κάνει συγκεκριμένες συστάσεις Είμαστε σε επαφή με την Κομισιόν η οποία κάνει προτάσεις για την ψηφιακή φορολογία και αυτό έχει μεγάλη σημασία και έτσι μπορούμε πάλι να επιβάλλουμε και να καταστήσουμε τον γενικό κανονισμό κάτι το οποίο θα έχει παγκόσμια και γενική ισχύ γιατί βεβαίως αφορά τον ψηφιακό κόσμο αλλά πάει και παραπέρα. Τώρα, οι δικές μου ερωτήσεις ε, προς τους ομιλητές είναι οι εξής ε, και προς εσάς. Ε. Γνωρίζοντας ότι ο κανονισμός αυτός ισχύει γενικώ και γνωρίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζουμε το τι συμβαίνει με τα δεδομένα των δικών μας πολιτών, τα οποία επεξεργάζονται πλατφόρμες σε ολόκληρο τον κόσμο. Όχι μόνο σε σχέση με την αγορά, όπου μπορεί να υπάρχει ένα σκάνδαλο σαν την Cambridge Analytica. Αν δούμε εταιρείε όπως η Huawei και η Alibaba, οι οποίες σύμφωνα με τον Κινέζο νομοθέτη πρέπει να αποθηκεύουν τα δεδομένα στην Κίνα. Για ποιο σκοπό, με ποιον τρόπο, τι θα κάνουμε εκεί. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αγνοούμε εμείς ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πολλά από τα κράτη μας έχουν συμβάσεις με αυτές τις εταιρείες για τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι ένα ερώτημα λοιπόν, πώς το έχετε σκεφτεί και τι μπορούμε να κάνουμε. Μετά, συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι αυτό απαιτεί εκπαίδευση των δικαστών, γιατί σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και θα έχουμε με την αυτή νομοθεσία πληθώρα τέτοιων υποθέσεων στα δικαστήρια, αλλά τι θα γίνει όταν οι χώρες, οι χώρες μας θα είναι υπεύθυνε Φανταστείτε ένα σκάνδαλο σαν αυτό το οποίο υπάρχει στην Ινδία τώρα με το πρόγραμμα Χαράρ, πώς λέγεται, ε, πρόγραμμα ταυτότητας, ε, ταυτοτήτων. Και οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι καταχρώνται τα δεδομένα των πολιτών για απάτες κτλ. Δηλαδή όταν το κράτος είναι υπεύθυνο για τις βάσεις δεδομένων ε, και γίνεται κατάξυση εκεί πέρα, ταυτοτήτων, φορολογικών στοιχείων κτλ. Και εκεί πέρα νομίζω μπορεί να βοηθήσει ο κανονισμός αυτός που περιέχει γενικούς κανόνες, ε, τους οποίους θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια βεβαίω. Αυτό το σκέφτονται οι εθνικές αρχές ε, όταν μιλάνε για την εφαρμογή του κανονισμού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να τελειώσουμε πρώτα με τους ευρωβουλευτές και μετά να ακούσουμε κάποιες τελευταίες απαντήσεις. Λοιπόν, η κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα συνάδελφοι. Ήδη ακούστηκαν διάφορα πράγματα, εγώ όμως θα ήθελα να επανέλθω στο ότι έχουμε πλέον έναν γενικό ευρωπαϊκό κανονισμό προστασία δεδομένων, αλλά πώς μπορούμε τελικά να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει ενιαία ερμηνεία. Γιατί ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 28, προσεχώς θα έχουμε 27 κράτη-μέλη που έχουν διαφορετικές αρχές προστασίας δεδομένων, μεγάλες χώρες, μικρές, με διαφορετικά μέσα στην διάθεσή τους. Οπότε τίθεται ένα ζήτημα ερμηνείας και ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου επόπτη εδώ. Θα ε, παρεμβαίνει όταν βλέπει ότι μια χώρα αποκλίνει στην ερμηνεία ή πηγαίνει προς μια λάθος πορεία, θα υπάρχει συνεργασία, θα ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές, προβλήματα ερμηνείας ε, θα μπορούν να συζητηθούν μεταξύ των αρχών. Θα παίξει ένα ρόλο και η Κομισιόν σε αυτήν την υπόθεση για να μπορέσει ακριβώς να οδηγήσει σε μία ενιαία εφαρμογή της ε, οδηγίας. Και βεβαίω υπάρχει και το ζήτημα των μικρών επιχειρήσεων αλλά και μη κερδοσκοπικών ε, οργανισμών. Τι θα κάνουν αυτοί, ειδικά στην περίπτωση στην οποία απαιτούνται ε, ακριβές ε, νομικές συμβουλές. Επίσης αναφέρθηκε το ζήτημα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και στις επιχειρήσεις. Αλλά υπάρχει και μια σημαντική ομάδα του πληθυσμού οι πιο ηλικιωμένοι, οι άτομα τα οποία υπεύθυνα και οι γονεί τους, οι γονείς επίσης που είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους και θα πρέπει να μπορούν ακριβώς να τα προστατεύσουν, να τα παρακολουθήσουν. Και όσον αφορά τώρα κάποιες πιο μεγάλες, συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις όπως το Facebook κτλ. θα πρέπει να δούμε εκεί πέρα πώς θα γίνει η εφαρμογή για να υπάρχει ακριβώς η προστασία των δεδομένων και μια συγκεκριμένη θα έλεγα περιχαράκωσή τους ε, τρόπων. την. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε άλλη μια βουλευτή, την κυρία Βίντε από την Ισπανία. Σας ευχαριστώ που με βάλατε τελευταία στιγμή στον κατάλογο των ομιλητών. Ο κανονισμός που αρχίζει να ισχύει σε 10 μέρες είναι μια κοινωνική αλλαγή που επηρεάζει το πρότυπο της εγγύησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη συμπεριφορά των φορέων, αλλά και τον τρόπο ελέγχου από τις ελεγκτικές αρχές. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή ε, είμαστε σε διαπραγμάτευση στο, στην, Κοινοβούλιο. Ε, έχουν ε, κατατεθεί πάνω από 350 τροπολογίες και θα, πρέπει, θα χρειαστεί να περιμένουμε να δούμε τι δουλειά θα κάνει η συγγήτρια για να αποβάλει σε αυτήν την ε, επιτροπή. Πιστεύω πως θα πρέπει ο κανονισμός να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα και γι' αυτό θα θέλω να ξέρω αν έχετε να μας κάνετε προτάσεις για τις χώρες που ήδη έχουν νομοθετήσει στον τομέα αυτό και έχουν ε, μακρά εμπειρία. Για μας θα χρησιμεύε για να προσπαθήσουμε να εντάξουμε αυτές τις προτάσεις στο κείμενο. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Ιντεφέλτ από την ομάδα ALDE του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ για την σημερινή συνεδρίαση, γιατί θυμάμαι τις πολλές ε, συνεδριάσεις που είχαμε για να καταλήξουμε σε αυτόν τον κανονισμό. Δουλεύαμε από το 2012, ουσιαστικά πριν τεθεί η πρόταση επιτάπητος. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει τόσο μεγάλη προσοχή για τον ε, κανονισμό και ευχαριστώ και την Cambridge Analytica που μας διαφήμισε τελικά. Αλλά αυτό το οποίο που μου προξενεί εντύπωση όπως και στους περισσότερους ομιλητές είναι ότι μας κάνουν ερωτήσεις άνθρωποι που ανησυχούν για το τι θα σημαίνει αυτός ο κανονισμός, εάν θα μπορούν να τον εφαρμόσουν ε, πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κόσμο εδώ πέρα ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν, όπως είπε η Μπίργκη Τσίπελ. Υπάρχει μια οδηγία που υπάρχει από το 1995. Και αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ότι προφανές, ε, το, ε, προφανές ότι το επίπεδο ενημέρωσης και η εφαρμογή του νόμου είναι τόσο χαμηλή ώστε ο κόσμος δεν ήξερε καν ότι υπήρχε ήδη προστασία δεδομένων. Δηλαδή αν κάποιο έχει μια εταιρεία σήμερα και τώρα συνειδητοποιεί ότι υπάρχει προστασία δεδομένων, τι έκανε τα τελευταία 20 χρόνια. Και αυτό πρέπει να μας ανησυχεί, γιατί ε, σαφώς δεν έχουμε κάνει την δουλειά μας. Όσον αφορά την ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις. Πολλοί κόσμος θεωρεί ότι είναι αναγκασμένος να συμμορφωθεί σε πολύπλοκες προδιαγραφές και μέτρα. Ενώ αυτά δεν αφορούν τους πάντες. Αν έχει κάποιος φούρνο, δεν τον αφορούν αυτά. Ή δεν είναι οι ίδιες προδιαγραφές με το Facebook. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να στείλουμε. Ε, μας χαλαρώσουμε, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Αυτό το οποίο με ανησυχεί και θα το συζητήσουμε το απόγευμα, αλλά δυστυχώ δεν θα είμαι εδώ, είναι η κατάσταση εφαρμογής ε, της οδηγίας. Ήταν πακέτο ρητός και λυπούμε για το ότι η εφαρμογή της οδηγίας είναι κοντά στο μηδέν. Τα κράτη-μέλη δεν βιάζονται καθόλου να την εφαρμόσουν. Γιατί? Και πραγματικά θα ήθελα να πω στους ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια να το θέσουν αυτό στα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί έχει περάσει ήδη η προθεσμία εφαρμογής. Νομίζω λοιπόν πως η Κομισιόν ε, πρέπει να το δει το ζήτημα και να φροντίσει τα κράτη-μέλη να την εφαρμόσουν οδηγία, αλλιώς να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Τελευταίος ερωτών, κύριος Μικολάσικ από την Πολωνία. Από την Εθνική Πολωνική Βουλή. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, όλα όσα είπατε για τους ανηλίκους, για τα παιδιά, μου φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά. Σημειώνονται πολλά προβλήματα ωστόσο και στην πράξη. Και εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι η γνώση γύρω από τον κανονισμό είναι περιορισμένη. Στην Πολωνική Γερουσία σχηματίσαμε μια ομάδα, εργασίας δηλαδή, για να εξετάσουμε θέματα προς των παιδιών στον επιγραμμικό κόσμο. Κυρίως μας απασχολεί η διαφάνεια στην προστασία των δεδομένων, κυρίως στην επεξεργασία των δεδομένων δηλαδή που κάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει να δίνουμε πληροφορίες κατανοητές και ιδίως όταν αυτές απευθύνονται σε ανηλίκους και σε παιδιά. Έχουμε τονίσει κατά επανάληψη ότι και οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν πώς θα μεταφέρουν το μήνυμα και στα παιδιά τους όταν τα παιδιά αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να γίνει επεξεργασία των δεδομένων τους και βεβαίως με όλα τα σχετικά προβλήματα. Εμείς γράψαμε και επιστολή στον Υπουργό Παιδείας της Πολωνικής Κυβερνήσεως και εν ώψη της επικείμενης εφαρμογής του GDPR και ζητήσαμε να οργανώσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και να τα περιλάβει και στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να γνωρίζουν τα παιδιά, να μάθουν τα παιδιά πώς προστατεύονται online. Χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση για τους ανηλίκους, για τα παιδιά βεβαίως ιδίως, αλλά και για τους δασκάλους, για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Και τονίζω με ιδιαίτερη ένταση το πόσο σημαντικό είναι να ενημερωθούν και τα πιο νεαρά παιδιά. Να βελτιώσουν τη γνώση τους για το πώς μπορούν να προστατεύονται, να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Και αυτό πρέπει να γίνει συστηματικά. Πρέπει να είναι, ξαναλέω, μια συνολική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Τελευταία, αλλά βεβαίω ε, εξίσου σημαντική με όλου του άλλου, η κυρία Χολμάιερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Ευχαριστώ. Βεβαίω, συχνά εμείς οι Γερμανοί διαβάζουμε τα όσα γράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έκανε ανακοίνωση τέλη Ιανουαρίου κατευθυντήριες γραμμές την λέει για την άμεση εφαρμογή του κανονισμού από την 25η Μαΐου. Βεβαίως, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, διάβασα μεν το έγγραφο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω περισσότερα από πριν. Όταν διαβάζω τώρα ότι η ειδική προστασία δεδομένων, δηλαδή ομάδα εργασία του άρθρου 29, μέχρι τώρα για θέματα όπως προφίλ, συγκατάθεση, διαφάνεια, πιστοποίηση, αναλογικότητα, δεσμευτικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, δεσμευτικότητα για την επεξεργασία, διατάξεις δηλαδή περί επεξεργασίας και όλα αυτά. Όταν βλέπω ότι όλες αυτές οι κατηγορίες γραμμές έως τώρα δεν υφίστανται, δεν έχουν εκδοθεί. Άρα, εμείς πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη προσπάθεια. Εμείς δηλαδή εδώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές στις χώρες μέλη, ώστε να υπάρχει κάποια ας πούμε ομοιογένεια στην εφαρμογή του κανονισμού. Δεύτερο, εάν θεωρήσουμε ότι οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είχαν εγκύψει το θέμα εδώ και πολλά χρόνια, και μιλούμε για τι μεγάλε επιχειρήσει επιχειρήσεις πρώτα-πρώτα. Για κοιτάξτε όμω τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε δεν έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν παροχή νομικών συμβουλών και πώς θα εφαρμόσουν αυτές τον κανονισμό. Έτσι λοιπόν δεν έχουν την απαραίτητη νομική παιδεία οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες και ούτε μπορούν, ξαναλέω, οικονομικά μιλώντας, να ζητήσουν την ε, παροχή νομικών συμβουλών. Άρα πρέπει το κράτος να τους βοηθήσει είτε μέσω των ε, εντεταλμένων την προστασία προσωπικών δεδομένων, εμείς όμως βλέπουμε στην Ομοσπονδιακή Γερμανία που είναι κράτος ε, ομοσπονδιακά δομημένο. Έχουμε 16 ε, κρατήδια και 16 διαφορετικές ερμηνείες του κανονισμού. Επομένως φανταστείτε τι θα γίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό τα βλέπω εγώ από κοντά κάθε μέρα. Θεωρώ ότι οι απλοί άνθρωποι έξω που τώρα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται περί πρόκειται. Δεν μπορούν να έχουν την ίδια αντίδραση όπως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουν την ανάγκη λοιπόν να τους δοθούν τα πράγματα έτοιμα, να μπορέσουν δηλαδή να τα κατανοήσουν. Είναι εύπεπτα. Και πρέπει βεβαίως, πρέπει να αντιληφθεί κανείς ότι υπάρχουν ήδη επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν τις ιστοσελίδες τους διότι φοβούνται ότι μπορεί να κάνουν κάποιο λάθος και να αρχίσουν οι καταγγελίες. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τις μικρές και εσεί επιχειρήσεις. Φανταστείτε την τελευταία μικρή επιχείρηση που διαθέτει μια ιστοσελίδα, ξαφνικά τρομάζει όμως, βλέπει του τίτλους τη εφημερίδα και λέει «Αμάν, θα αρχίσουν οι καταγγελίες». Πρέπει να αντιληφθεί λοιπόν και το ανώτατο επίπεδο ότι οι απλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν όλες αυτές ε, τις ε, υψηλές απαιτήσει. Πρέπει λοιπόν να τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται και όχι να ερχόμεθα άνωθεν να δίνουμε μόνο μαθήματα καλής διαγωγής. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα επανέλθω τώρα στα μέλη του πάνελ και θα τις παρακαλέσω να απαντήσουν σε οποιασδήποτε ερωτήσεις, σε επιθυμούν. Η κυρία Γέλνεκ πρώτη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις διάφορες ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στο πρόσωπό μου. Πρώτα στην ερώτηση της κυρία Γκόμες σχετικά δηλαδή με το εάν φέρει την ευθύνη το κράτος. Δεν αποκλείονται, δεν εξαιρούνται οι κρατικές αρχές από την εφαρμογή των προτύπων και οι αρχές προστασίας δεδομένων έχουν το καθήκον να παρακολουθούν την τήρηση και την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και θα πρέπει να το πράξουν αυτό και να το εφαρμόζουν και στις εθνικές αρχές. Δεύτερο έγινε το ερώτημα της ε, ερμηνείας, της κοινή ερμηνείας, δηλαδή σχετικά με μικρές και μεγάλες αρχές προστασίας δεδομένων και ποιο ρόλο παίζει ο Ευρωπαίος εντεταλμένο στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και αν γίνεται κάποια ανταλλαγή απόψεων και ποιο είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως και ήδη προετοιμάζουμε την δυνατότητα να υπάρχει μια όσο το δυνατόν πιο συνεκτική ερμηνεία των διατάξεων του κανονισμού. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό στο μέλλον όλο και περισσότερο. Οφείλουμε να το κάνουμε. Γνωρίζετε ότι υπάρχει και Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων η οποία καλείται να φροντίσει ώστε ο κανονισμός να εφαρμόζεται ομοιογενώς σε όλες τις χώρες μέλη. Η δε συνεργασία με τον Ευρωπαίο εντεταλμένο την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επίσης καθήκον των αρχών προστασίας δεδομένων. Δηλαδή, αποτελεί και αυτός μέρος της ομάδας των αρχών προστασίας δεδομένων. Δεν ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζεται από τον κανονισμό. Μπορεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από την Επιτροπή Προστασία Δεδομένων να γνωμοδοτεί για ορισμένα θέματα και να τοποθετείται. Θέματα δηλαδή τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τίθεται το ερώτημα μετά οι μικρέ οργανώσει. Πώ μπορούν να υποστηριχτούν. Εξ όσων ξέρω, όλε οι αρχέ προστασία δεδομένων στην Ευρώπη έχουν ήδη περιλάβει στι ιστοσελίδε του πολλά πράγματα. Παίρνω παράδειγμα τη δική μα, την Αυστριακή. Έχουμε guidelines για μη νομομαθής και μάλιστα εκεί γίνονται πάρα πολλές ερωτήσεις από το κοινό και εκεί έχουμε περιλάβει και ερωτηματολόγιο που μπορούν να εξετάζουν δηλαδή οι χρήστες να δουν α, ποιο από αυτά τα πράγματα με αφορά και ποιο, και ποιο όχι. Και ξαναλέω είναι για μη νομομαθείς. Έχουμε και ένα newsletter το οποίο φροντίζουμε ώστε να είναι απολύτως κατανοητό ώστε να μην χρησιμοποιείται δηλαδή αυτή η ειδική γλώσσα των νομικών. Και αυτό ε, για όλες τις ε, νομικές διατάξεις. Τώρα, οι εκπαιδεύσεις. Οι γονείς που πρέπει να παρακολουθούν το τι κάνουν τα παιδιά τους. Νομίζω ότι όσοι έχουν μικρά παιδιά δεν είναι παραπάνω το πολύ πολύ από 50 ετών και άρα γνωρίζουν να χειρίζονται το διαδίκτυο. Τι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί οι οποίοι, επιχειρήσεις που δεν έχουν φροντίσει να τηρήσουν τα της προστασία δεδομένων και ξύπνησαν όταν ξαφνικά τους επευλήθη κάποια ποινή. Και μάλιστα και οι ανώτατοι υπευθυνοί τους υπέστησαν κυρώσεις. Όσοι τήρησαν βέβαια τις διατάξεις του νόμου δεν έχουν πέσει, ε, δεν έχουν δηλαδή ε, δεν τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Θα πρέπει βέβαια αυτά να γίνουν ορατά. Ιδίω για αυτούς οι οποίοι δεν τηρούν τις διατάξεις του νόμου. Αυτό δεν μπορεί βέβαια να είναι καθήκον της αρχής προστασίας δεδομένων. Είναι κοινωνικό καθήκον. Βεβαίως, τι, σε εσά τα λέω, εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά ως ευρωβουλευτές. Τελευταίο, η, εκπο... Ε, από τη Γερμανία. Οι guidelines της ε, Επιτροπή του άρθρου 29, τη ομάδα τη έργασια του, άρθρου 29. Υπάρχουν ε, σχετικές κατευθυντήριε γραμμές, οι οποίε δημοσιεύονται, κάποιο διακόπτει από κάτω χωρίς μικρόφωνο, η κυρία Τώρα μόλις μπήκαν στην ιστοσελίδα. Μέχρι τώρα, ε, σύμφωνα, με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπήκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου. Εκτό αν λέει κάτι λάθο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, όχι, βεβαίω δεν σα αντιμιλώ. Γνωρίζω όμω από ιδίαν εμπειρία ότι αυτέ οι κατευθύνε γραμμέ βρίσκονται στην ιστοσελίδα τη ομάδα εργασία 29 από μακρότερου χρονικού διαστήματο. Ανεξαρτήτω του πότε εγκρίθηκαν. Πάντω το τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, η παρέμβασή σα για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Βεβαίω κατανοώ τι λέτε τα επιχειρήματά σα. Όμω, ο φόβο που έχουν ορισμένες μικρές και μεσές επιχειρήσει δεν οφείλεται στις διατάξεις του βασικού κανονισμού. Υπάρχουν πολλέ οργανώσεις που εκπροσωπούν επαγγελματικά συμφέροντα, επαγγελματικέ οργανώσεις κλπ. Και εκεί βεβαίω είναι υποχρεωτικά μέλη οι, διάφορες, ε, τα, διάφοροι επαγγελματίες. Έχουν οργανώσει ε, ενημέρωση των μελών τους. Ε, για ορισμένους δεν ήταν επαρκές αυτό. Για τον ε, βασικό κανονισμό πάντως υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, υπάρχουν πολλοί μάλλον που φοβίζουν τις μικρές επιχειρήσεις, λέγοντάς ότι θα υποστούν βαρύδα τις κυρώσεις, κάτι το οποίο όμως δεν είναι ορθό. Όλοι πρώτα θα προειδοποιούνται πριν να υφίστανται κυρώσεις. Βεβαίως λαμβάνονται υπόψη όλα μέσα σε ένα πλαίσιο αναλογικότητας. Βεβαίως και ο Κρεοπόλης και και ο, και και ο Φούρναρης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να γνωρίζουν. Αλλά δεν έχουν βεβαίως τις ίδιες ευθύνες με τον κύριο Μάρκ Ζούκερμπεργκ του Facebook. Ευχαριστώ κυρία Γέλινεκ. Ακολουθεί η κυρία Τζιμέλοβιτς. Ευχαριστώ. Έχω να κάνω πάρα πολλέ παρατηρήσει, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω για τι πιο σημαντικέ σε σχέση με το κανονισμό αντιτράστη για τι πλατφόρμε. Είναι η επόμενη μεγάλη μάχη και ελπίζω πω θα συμβεί και εδώ, ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την αυτό το θέμα. Αν και θέλω να κάνω έκκληση στα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου να θυμηθούν ότι δεν θέλουμε να διχάσουμε τι εταιρείε, δεν θέλουμε να διχάσουμε τι πλατφόρμε αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε είναι να δούμε τη διαλειτουργικότητα και να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε την πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες χωρίς να τους καταστρέψουμε, ώστε να υπάρχουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες και έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να τις χρησιμοποιεί, αλλά με ε, υψηλότερες κανόνες ε, προστασίας. Αυτό είναι το σχόλιο μου προς την κυρία Κόμες. Το στηρίζω αυτό που είπατε. Ε, τώρα, πολλά σχόλια πιστεύω πως κινούνται από το φόβο πως οι μικροί οργανισμοί, μικρές επιχειρήσεις θα υποφέρουν από τον κανονισμό αυτό ή επειδή δεν ενημερώνονται σωστά. Συμφωνώ με τον κύριο, την κυρία Σελινέκ ότι υπάρχουν ε, διάφοροι πόροι ε, ε Υπάρχουν ε, μη κυβερνητικοί οργανισμοί με πολλές γνώσεις, ε, όμως δεν έχει γίνει μια ισχυρή δημόσια εκστρατεία, κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ως ΜΚΟ. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια ως ομάδες ε, ΜΚΟ από διάφορες χώρες προσπαθήσαμε να κάνουμε έκκληση στην, στα ευρωπαϊκά μέσα και όργανα και διαρκώς ακούμε ένα μεγάλο όχι. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό. Πιστεύω πως είναι πολύ κακό κακό γιατί γιατί από την πλευρά των όσων έχουν προπολογισμό για αυτήν, αυτού του είδους τις δραστηριότητες να μην στηρίζουν ε, για την ενημέρωση. Είναι μεγάλο λάθος ε, και τώρα το πληρώνουμε ε, γιατί ε, έχει αναπτυχθεί πολύ παραπληροφόρηση σε σχέση με τον νέο κανονισμό. Τέλος, για τα όσα κυρία Ιντβέλτε, συμφωνώ ότι είναι μεγάλη πρόκληση η εφαρμογή του πακέτου και μπορώ να σας δώσω παραδείγματα από τη χώρα μου γιατί στην Πολωνία η εφαρμογή της οδηγίας δημοσιεύθηκε μόλι πριν δύο εβδομάδες. Είναι ακόμα νομοσχέδιο, δεν έχει υιοθετηθεί. Και έχει τόσε πολλέ εξαιρέσει που έρχεται τελικά σε αντίθεση με τη λογική της οδηγίας. Δηλαδή θα έχουμε χαμηλότερε ε, διαγραφές αν αυτό εγκριθεί, εάν ε, από ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής και εξαίρεση ε, πλήρης για όλες τις αρχές αρμόδιες για την επιβολή του νόμου ή για, οτιδήποτε έχει να κάνει με πληροφορία ξερούνται πλήρως και η πρόσβαση ε, για τους πολίτες δεν θα υπάρχει. Ε, θα πάει πάρα πολύ κακά λοιπόν αυτό το πράγμα, πολύ άσχημα και φοβούμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσει να εμποδίσει αυτή την κατάσταση. Αν δούμε την εξαίρεση για τη δημόσιο τομέα, αυτό έχει ήδη προβλεφθεί από τα κρατημέλη. Ε, και θα πρέπει καλύτερα να το ελέγξει και να το παρακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, τέλος, περνάμε στην κυρία Ένιον. Έχετε τον λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαπιστώνω ότι έχουμε πάρα πολλές, εκείνες κοινέ ανησυχίες. Δηλαδή στις επόμενους μήνες και χρόνια θα, συνεχίσουμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα, ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο για θέματα που είναι τόσο θεμελιώδη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο συντονισμού να παίξει ανάμεσα σε όλες τις εθνικές αρχές ώστε να εξασφαλίσει πως οι ερμηνείες θα είναι οι ίδιες και ότι θα τεθούν σωστά σε εφαρμογή. Ε, για να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα σε σχέση με τις μικρές ε, ε, εταιρείε. Αυτό το μήνυμα που θέλουμε εμείς να στείλουμε είναι μια από τις αρχές που περιλαμβάνονται στο νέο κανονισμό και που είναι κάτι το νέο, όλα βασίζονται στην, ανάλυση κινδύνου. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση ένας ε, φούρναρης με το facebook φυσικά ε, και αυτό θα πρέπει σωστά να μεταβιβάζεται και να γίνεται κατανοητό. Και πάλι οι καλές πρακτικές που θα πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ μας και ε, στο πλαίσιο των αρμόδιων αρχών. Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας που θα πρέπει να συνεχιστεί και να συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε. Να εξασφαλίζουμε ότι είμαστε στη σωστή καμπύλη προόδου και εάν έχω μια ευχή να εκφράσω σε σχέση με τα όσα άκουσα και σε σχέση με τους φόβους που εκφράζονται από την ε, παρακαθήμενή μου, ε, θα ήταν δυνατόν να έχουμε μία σύγκριση όλων αυτών των κειμένων. Ε, θα μπορούσε αυτό να γίνει από την Κομισιόν, αλλά και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να δεσμευθεί σε αυτή την πορεία, ώστε να δούμε ακριβώς ποια είναι τα σημεία που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να υπάρξει καλύτερη σύγκληση στα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ. πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας σε αυτήν την συζήτηση. Ευχαριστώ τις ομιλήτριες. Η κυρία Γέλνεκ έφυγε ήδη. Τώρα προσκαλέσω τους ομιλητές του δεύτερου μέρους. Τον κύριο Ζουντίκα Ελφάν, τον κύριο Λουκ Έντριξ ε, και την κυρία Πασκάλ Γκέλη και το δεύτερο τμήμα επίσης αφορά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού σε σχέση με τον αντίκτυπο που έχει στον ιδιωτικό τομέα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήδη μας απασχόλησαν και τώρα θα μπορέσουμε να επεκταθούμε. Πρέπει λοιπόν, να σας παρακαλώ. Okay, uh, Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ξεκινάμε σήμερα με το δεύτερο τμήμα της ε, συζήτησής μας για την εφαρμογή του πακέτου προστασίας δεδομένων. Στο δεύτερο τμήμα λοιπόν καλωσορίζω στο βήμα τον κύριο Ζουτικά Ελφάν, αναπληρωτή διευθυντή της νομικής υπηρεσίας της Ubisoft, τον κύριο Λουκ Εντρίξ, διευθυντή ε, επιχειρησιακής πολιτικής ε, της Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την κυρία Πασκάλ Γκαλή, η οποία είναι αρμόδια προστασίας δεδομένων του ομίλου Schneider Electric. Σας καλωσορίζω λοιπόν και αμέσως δίνω τον λόγο στον πρώτο μας ομιλητή να σας υπενθυμίσω πως τώρα είναι κίτρινα τα χαρτάκια που συμπληρώνετε για να ζητήσετε τον λόγο και οι ευρωβουλευτές ως συνήθως μπορούν να μου κάνουν νόημα. Λοιπόν, τον λόγο έχει ο κύριος Ελφάν για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. Εξ ονόματος της Ubisoft είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το θέμα που αφορά την προστασία των δεδομένων. Όπως γνωρίζετε αυτή η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία περιλαμβάνει ε, αξίε ε, που είναι γεννή δημοκρατία δημοκρατίας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων αλλά και την προστασία τη ιδιωτική σφαίρα, ιδιωτική ζωή, προσωπικής ζωής. βλέπουμε την άφηξη αυτού του κανονισμού ως ευκαιρία και ατού για τους ε, πολίτες, τα, τα, τα πρόσωπα. Η θετική πτυχή αυτού του κανονισμού είναι ότι φωτίζεται η Ευρώπη των προσωπικών δεδομένων, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής για τα προσωπικά δεδομένα και χάρη σε αυτό το κανονισμό βλέπουμε ότι όλα ένα και περισσότερο υπάρχει μια ομοιογένεια των προσεγγίσεων για τα προσωπικά δεδομένα στην Ευρώπη. Έχουμε περισσότερο μια προσέγγιση εντό Ευρώπης ε, ότι δηλαδή πρόκειται για μια αξία ενώ ε, στην Αμερική φαίνεται τα δεδομένα να θεωρούνται ως κάτι το άειλο ε, και γι' αυτό και είμαστε ευχαριστημένοι που στην Ευρώπη έχουμε ε, ε, στόχο περισσότερη προστασία. γιατί την Ubisoft είναι μια εταιρεία που προτείνει παιχνίδια βίντεο. Υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Έχουμε 13.000 κόσμο, ασχολούνται σε, σε, σε, στις 5 υπήρους. Είναι εγκατεστημένοι και έχουμε 500 εκατομμύρια παίκτες και τους προτείνουμε ε, ε, διαδραστικά παιχνίδια είτε σε κονσόλα, είτε σε κινητό, είτε στην τηλεόραση και για να επιτύχουμε την εμπιστοσύνη των παικτών πρέπει να σεβόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα και γι' αυτό και θεωρούμε ότι αυτός ο κανονισμός είναι μια ευκαιρία να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των παικτών γιατί αν θέλει κανείς να δημιουργήσει παιχνίδια βίντεο για να βγάλει τον ιό πούμε όταν ε, υπάρχει πρόβλημα ή για να δημιουργήσει νέους κόσμους, νέες ιστορίες χρειάζεται τα προσωπικά στοιχεία. Είναι αυτό απαραίτητο και γι' αυτό και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ε, αυτός ο κανονισμός μας προσφέρει περισσότερα μέσα ελέγχου και ευκαιρίες ε, ταυτόχρονα. Ενισχύεται η φήμη μας επίσης. Είναι μια ευκαιρία για να ενισχύσουμε την διακυβέρνηση των στοιχείων μας με χαρτογραφικά στοιχεία και να μετατρέψουμε τις νομικές ε, υποχρεώσεις σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ε, έχουμε φτιάξει λοιπόν διάφορες δράσεις, έχουμε ενισχύσει την ομάδα μας που είναι ε, αρμόδια για τα στοιχεία, έχουμε χαρτογραφήσει τα στοιχεία μας, έχουμε φτιάξει ένα εργαλείο ώστε να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια και έλεγχος όπως για τους παίχτες μας και έχουμε φτιάξει και μια εσωτερική ομάδα εργασία. Όσον αφορά την ενίσχυση των ομάδων μα, έχουμε ενισχύσει τι ομάδε μα σε θέματα ε, στοιχείων και προστασία. Έχουμε αυτή την ευκαιρία, αλλά όπω είπατε, ε, ε, δεν είναι αυτό το ίδιο για πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει και Ξέρουμε ότι είναι πιο περίπλοκο. Έχουμε δημιουργήσει ε, άτυπες ομάδες εργασίας στο πλαίσιο της Ubisoft που συνεδριάζουν κάθε μερινά αλλά και κάθε εβδομάδα ώστε να δημιουργηθούν ε, σε δεσμοί και ε, εσωτερικές επαφές ώστε να προτείνουμε μέσα ελέγχου σε όλους τους παίκτες. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και θα αναπτυχθεί τους επόμενους μήνες. Η ιδέα είναι να ενημερωθεί και το e-privacy γιατί πεδράσαμε από ε, οδηγία σε κανονισμό. Το λυπούμεθα που το e-privacy δεν υιοθετήθηκε ταυτόχρονα με το κανονισμό αυτό. Προβλέπουμε ε, κάπως, προσπαθούμε μάλλον να δούμε τι γίνεται με το e-privacy αλλά δεν μπορούμε και προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο για την ιδιωτική ζωή για να έχουμε την εμπιστοσύνη των παικτών και να αποφύγουμε σκάνδαλα. Επίσης χαρτογραφήσαμε τα στοιχεία μας ε, αλλά αυτό γίνεται παντού ε, για σας, για τους, για τους υπολογιστές σας, για το mail σας. Υπάρχουν στοιχεία που υπάρχουν παντού και έχουμε εταίρου που μας λένε ε, αυτή τη στιγμή είμαστε ικανοποιημένοι που έρχεστε με ενισχύσει στα θέματα της ιδιωτική ζωής γιατί εμεί είχαμε αμφιβολίες. Σήμερα επειδή είναι όλα χαρτογραφημένα έχουμε καλύτερες δυνατότητες διακυβέρνηση των στοιχείων. Αυτό είναι μάλιστα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πλεονέκτημα για να φτιάξουμε καλύτερα παιχνίδια. Ε, τεράστιο πλεονάκτημα, ε, η χαρτογράφηση των στοιχείων που μας επιτρέψει είναι επίσης να συζητήσουμε με όλους μας τους συνεργάτες και να ευαισθητοποιήσουμε στο θέμα της ιδιωτικής ζωής και να τους εξηγήσουμε ότι χάρη στο νέο κανονισμό όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν να σας εντοπίσουμε έμεσα ή άμεσα όπως τα cookies ας πούμε είναι στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και εδώ έχουμε ένα, μια αναλλαγή νοοτροπίας να τους εξηγήσουμε ότι υπάρχει και θέμα ε, όταν υπάρχουν στοιχεία στοιχεία ενός παίκτη που συνδέονται με ένα τεχνικό ε, στοιχείο αναγνώρισης και αυτή είναι μια επανάσταση ε, σε θέματα νοοτροπίας και πρέπει να το συζητήσουμε με όλους ε, που, τους εμπλεκόμενους και θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλους μας τους συνεργάτες να προχωρήσουμε και στο σχεδιασμό να, σχεδια... να ευαισθητοποιήσουμε 13.000 κόσμο που εργάζεται για μας ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε online μια ομάδα που μας επιτρέπει να έχουμε... Έχουμε παιχνίδια όπως το Assassin's Creed, ε, όπως το James Dance και παιχνίδια που, ας πούμε, θα τα χρησιμοποιήσουμε τους χαρακτήρες σε συμπαθητικά και ευχάριστα βίντεο, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους συνεργάτες μας και τους παίκτες. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, που δεν έχουν τα μέσα να φτιάξουν τέτοιο είδους ε, βίντεο. Ίσως οι αρχές προστασίας των δεδομένων θα μπορούσαν να φτιάξουν, να σκεφτούν και να φτιάξουν και να ευαισθητοποιήσουν ε, τον κόσμο εκείνες. Επίσης ενισχύουμε την ασφάλεια των βασιών ε, δεδομένων μας, ε, γιατί καθημερινά προσπαθούν οι hacker να μπουν σε αυτές. Έχουμε πάνω από 1.500 υπαλλήλου που ασχολούνται με αυτό την υπόθεση και προσπαθούμε να φτιάξουμε ειδικευμένε ομάδες ε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε κάθε πιθανότητα ρήξη της ασφάλειάς μας. Έχουμε ομάδες που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο και είναι επίσης η ευκαιρία για να ενισχύσουμε την νομική μας ασφάλεια, τις υποχρεώσεις μας που απαιτούμε και από πλευράς των συνεργατών μας προσπαθούμε να, εμπνεώσουμε, να, να εμπνευτούμε από τα όσα προτείνει η ΚΝΙΛ, η Γαλλική Αρχή, όσον αφορά το, την, προστασία των δεδομένων και βλέπουμε το εύρος του κανονισμού μας ε, ε, γιατί οι Αμερικανοί εταίροι μας προσπαθούν να μας πιέσουν. Εμείς προσπαθούμε να πιέσουμε με βάση αυτόν τον κανονισμό που θεωρούμε πως είναι καθολικός. Είναι θετικό αυτό το στοιχείο. Είναι επίσης λιγότερα τα τυπικά ε, βήματα προς τον αρμόδιο ρυθμιστή αναλαμβάνει ευθύνη βέβαια η εταιρεία, αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, και μπορέσαμε, είχαμε κάποια εμπόδια Όσον αφορά την εξοεδαφικότητα, ε, τέθη το θέμα του κατά πόσο πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός σε όλους τους παίκτες. Ας πούμε, σε έναν Κινέζο παίκτη θα του επιβάλλουμε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και αν έρθει στην Ευρώπη υπόκειται στον κανονισμό. Είπαμε ότι εμεί θα εφαρμόσουμε αυτό, τους ίδιους κανόνες σε όλους τους παίκτε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί αυτό μας επιτρέπει να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη από τους παίκτες και τους ανθρώπους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προτείνει η Ubisoft. Είπαμε λοιπόν θα εφαρμόσουμε τους ίδιους κανόνες για όλους. Έπειτα έχουμε περισσότερα αιτήματα ε, για συμμετοχή, για πρόσβαση κάποιες φορές υπάρχει μόνο ένας τεχνικός ε, τύπος αναγνώρισης. Δεν έχουμε καν το όνομα του ατόμου, του ανθρώπου, δεν έχουμε καν το email του. Ε, αυτά τα ερωτήματα τα θέτουμε στον ρυθμιστή είναι ζητήματα που βλέπουμε πολύ τακτικά και για, πρέπει να έχουμε ε, κοινή προσέγγιση και συνεργαζόμαστε με επαγγελματικού ε, ε, και ενώσει, με την ίση την SNGV όσον αφορά τα βιντεοπαιχνίδια. Και μία τελευταία παρατήρηση χρειάζεται να έχουμε μία <laughs> ομοιογενή προσέγγιση στην εφαρμογή του κανονισμού. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων να μην έχει ε, ε, αρκετό βάρος και κύρος, γιατί αυτό σημαίνει διαφορές ανάμεσα στις αρχές προστασίας των δεδομένων, ανάμεσα στις θέσεις που υιοθετήσουν, πράγμα που ήδη έχει συμβεί. Ε, αυτή είναι η πραγματική δυσκολία. Και έπειτα, όταν θα υιοθετηθούν μέτρα, πράξεις, προσπαθήστε να είστε όσο γίνεται πιο ομοιόμορφοι, ομοιογενείς, να αποφύγουμε επιπλοκές και εμπόδια. Γιατί ο στόχος του κανονισμού είναι κοινή να είναι κοινό. Εμείς βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον κανονισμό ως μια ευκαιρία ε, εμπιστοσύνη και ανάπτυξης και είναι κάτι ε, όπου πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε ο κόσμος που είναι όλο ένα και πιο ψηφιακός να σέβεται τους χρήστες Το Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαν. Θα ακολουθήσει ο κύριος Χέντριξ. Έχετε το λόγο κύριε, 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν φαίνεται η παρουσίασή μου. Ωραία, σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που μας ε, καλέσατε σήμερα εδώ και ενδιαφέρον είναι και ο τίτλος ε, «Η επίπτωση στον ιδιωτικό τομέα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Μην ξεχνάμε ότι 99,8% των επιχειρήσεων είναι μικρές και μεσαίες. Και πάλι λοιπόν σας ευχαριστώ που μας καλέσατε για να μας ακούσετε. Όσοι δεν είναι εντός της φούσκας των Βρυξελών ίσως να μην ξέρουν την ΟΕΑΠΜΕ. Πρόκειται για την οργάνωση των εργοδοτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή εκπροσωπούμε τις εθνικές ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε 67 ενώσεις μέλη, εθνικές και κλαδικές ευρωπαϊκές. Συνολικά εκπροσωπούμε 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε 24 χώρες, μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μην πω μικρές και μικροσκοπικές θα ήθελα να επανέλθω στο 2012. Ε, είχαμε επίσης ανύποπτο χρόνο. Μπορείτε να τα δείτε αυτά στην ε, σελίδα μας όταν είχαμε κάποιες προσδοκίες για τον νέο κανονισμό και μπορείτε να δείτε εάν τα όσα ζητούσαμε τότε ε, επιτέχθησαν. Πρώτα απ' όλα είναι σαφές αυτό ότι έπρεπε να λάβουμε υπόψη τις νέες ε, τεχνολογικές εξελίξεις, ε, ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, αυτό οπωσδήποτε το πετύχαμε, αλλά και μια ισορροπημένη προσέγγιση και να αποφύγουμε το υπερβολικό διοικητικό βάρος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ανάγκη για ξεκάθαρα και σαφώς διατυπωμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ε, εδώ πέρα, ε, για να μην έχουμε μεγάλα προβλήματα και να μην υπάρχει επιπλέον διοικητικό βάρος για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, να έχουμε διατάξεις οι οποίες θα είναι κατανοητές και φιλικές προς τον χρήστη. Και το τελευταίο το οποίο αναφέρθηκε και στο προηγούμενο πάνελ εκστρατείες ενημέρωσης ε, για τα προσωπικά δεδομένα με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τους, ε, τις οργανώσεις ε, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτά τα είχαμε πει το 2012 ερχόμενοι τώρα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, και τον γενικό κανονισμό, θα ήθελα να τονίσω πρώτα απ' όλα ότι πρώτα απ' όλα εμείς ως επιχειρηματίες ενδιαφερόμαστε πολύ για την ιδιωτικότητα την δική μας και των ε, πέλατων μας και επίσης ενδιαφερόμαστε ε, βεβαίω για το κράτος δικαίου. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, πρέπει να σέβονται την νομοθεσία. Και τότε είχαμε υποδεχτεί θετικά την πρόταση της Κομισιόν, την οποία βρήκαμε πολύ ισορροπημένη και είχε ακριβώς την πρόθεση να υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το τελικό κείμενο μπορούμε να πούμε ότι δεν σέβεται την προσέγγιση ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα τον μικρό και η απόδειξη είναι απλή. Ο νόμος ονομάστηκε Lex Google, δηλαδή ε, κυρίως αφορούσε τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τις μικρές και τις μεσαίες. Ε, παρ' όλα αυτά εμείς ζητήσαμε να ενσωματωθούν και τα δικά μας τα σχόλια. Τέλος πάντων, αυτά έγιναν. Τι κάναμε λοιπόν οι οργανώσεις μας ε, στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αφιέρωσαν πολύ χρόνο στην ενημέρωση και στο να αναπτύξουμε εργαλεία για τις μικρές ε, και μεσαίες επιχειρήσεις ε, στο εθνικό και στο κλαδικό επίπεδο, γιατί ο κάθε κλάδος χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση και αυτό νομίζω συμφωνεί και με το εκτιμώντας την αιτιολογική σκέψη 132 του κανονισμού που μιλάει για το ότι επαφίεται στους εθνικούς επόπτες η παροχή πληροφοριών, αλλά ήταν κάτι το οποίο ανέλαβαν οι δικές μας οργανώσεις. Επίσης, στο εθνικό επίπεδο υπήρχε πολλή συνεργασία με τους επόπτες προσωπικών δεδομένων, πολύ καλή συνεργασία, χωρίς να είναι παντού ιδεώδης, αλλά τελικά νομίζω ότι τώρα σε όλες τις χώρες υπάρχει μια καλή συναντήληψη μεταξύ των επιχειρηματικών ενώσεων και των εποπτών προσωπικών δεδομένων και οπωσδήποτε θα αναπτυχθεί τις επόμενους μήνες. Όλα αυτά όμως σημαίνουν και μεγάλο κόστος και αβεβαιότητα και θα επανέλθω σε αυτό και κατακαιρματισμό και διαφορές και δυσκολίες στην εφαρμογή του κανονισμού και βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει μια έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού για κάποιες θέσεις και υπάρχει και η δυσκολία της ε, μη κατανόησης της νομοθεσίας. Θα σας δείξω κάποια δεδομένα, το τι πρέπει να διαβάσει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον κανονισμό που είναι 88 σελίδες στην επίσημη εφημερίδα της ε, κοινότητας, ε, σχεδόν 100 άρθρα η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 δημοσίευσε 9 κατευθυντήριε γραμμές, ε, πέντε από αυτές μετά από τον Ιανουάριο του 18, η τελευταία 16 Απριλίου του 18, που ήταν πάρα πολύ σημαντική και αφορούσε την συνένεση. Συνολικά 237 σελίδες. 158 σελίδες φέτος. Το 60% δηλαδή δημοσιεύτηκε μόλις φέτος. Και η πιο τέσσερις πιο πρόσφατες είναι ακόμα μόνο στα αγγλικά, το 70%. Και εκεί πέρα έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί ε, εγώ είχα την εντύπωση ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε γενικές γραμμές πρέπει να επικοινωνούν στην γλώσσα του πολίτη. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, το Κοινοβούλιο έλαβε υπόψη τις μικρόμεσες επιχειρήσεις στο άρθρο 30 εδάφιο 5 λέει ότι ε, οι υποχρεώσει αυτέ ε, στι παραγράφου 1 και 2 δεν θα ισχύουν σε μια επιχείρηση που απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και μετά ξεκινούν οι εξαιρέσει. Εκτό εάν η επεξεργασία αυτή δεν είναι ε, συγκυριακή. Ε, απευθυνθήκαμε λοιπόν στην Επιτροπή και λέμε πώ το ερμηνεύεται αυτό. Γιατί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν δεχτεί ένα κείμενο που έλεγε οι μικρομεσαίε επιχειρήσει εξαιρούνται. Αλλά η ομάδα εργασία του άρθρου 29 δεν μα έχει ακόμα απαντήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια απάντηση στη σελίδα του. Στην γνωμοδότηση της 16ης Απριλίου λέει όχι έχουμε μια αυστηρή ερμηνεία γιατί κάθε εταιρεία στην πραγματικότητα ε, επεξεργάζεται δεδομένα ε, τακτικά. Οπότε δεν εξαιρούνται οι μικρόμεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε δεν ισχύει αυτό το άρθρο. Δεύτερον, ανέλαβε υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Κοινοβούλιο το ανέφερα, ήδη στο εκτιμώντας 13 λέγεται ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των ε, μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ε, ναι, έχουμε το άρθρο 35, αλλά όπως σας είπα ήδη δεν πρόκειται περί εξαίρεσης. Αλλά τα κράτη-μέλη και οι επόπτες δεδομένων ενθαρρύνονται και ελπίζουμε να γίνει αυτό να ληφθούν υπόψη οι ειδικέ ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην εφαρμογή του κανονισμού μετά την 25η Μαρτίου και μετά θα σας, δώσω την, ε, θα σας δείξω τη σελίδα τους. Ε, δεν έχω τώρα σκοπό εδώ πέρα να κατηγορήσω κάποιον. Βλέπετε εδώ πέρα την σελίδα της ε, Βελγικής Εποπτικής Αρχής επειδή είμαι Βέλγος για να μην κατηγορήσω κάποια άλλη χώρα. δεν κατηγορώ δηλαδή. Είναι απλά ειλικρινής. Αν διαβάσετε το τι λέει, λέει το εξής. δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό είναι στις συχνές τους ερωτήσεις. Γιατί δεν μπορούμε ακόμα να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας. Και στην επόμενη σελίδα λέει, ε, δίνει κάποιες ε, περισσότερες εξηγήσει. Αυτή είναι η κατάσταση στις 23 Απριλίου πριν από λίγες μέρες. Γιατί δεν μπορεί η Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις μας. Γιατί είναι ένα έργο εν εξελίξη και δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς θα οριστικοποιηθεί. Αυτά μας τα λένε οι επόπτες προσωπικών δεδομένων. Οπότε η μόνη ε, λύση ε, λοιπόν που μας απέμενε ήταν ε, να απευθύνουμε μια επιστολή μαζί με την Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στην Επίτροπο την κυρία Γιούροβα ζητώντας μία περίοδο χάριτος ενός έτους για να συσταθεί στα κράτη-μέλη και στις εθνικές εποπτικές αρχές να επενδύσουν περισσότερο στην συμβουλή και στην στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να δεσμευτούν ότι στα πρώτα χρόνια δεν θα επιβάλλουν πρόστιμα αλλά θα κάνουν μόνο συστάσεις σε περίπτωση ε, παραβάσεων. Νομίζω αυτή είναι η προσέγγιση, δηλαδή να γίνουν κάποιες συστάσεις για να λυθούν πρώτα τα προβλήματα. Και πρέπει να πω ότι σε πολλές χώρες ε, το ίδιο έχουν κάνει οι οργανώσεις μέλη μας. Έχουν ζητήσει δηλαδή από τα κράτη τους ε, μία τέτοια περίοδο χάριτος. Νομίζω τελείωσε και ο χρόνος μου. Να πω μόνο το εξή. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να μας βοηθήσουν σε αυτό το αίτημα για μια περίοδο χάριτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εγώ. Ακολουθεί η κυρία Γκελή. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμες και αξιότιμοι ευρωβουλευτές και βουλευτές εθνικών βουλών. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών που μου δίνετε την ευκαιρία να σας εξηγήσουμε το πρόγραμμα της ε, οργάνωσης που εκπροσωπώ και τι από αυτά λειτουργεί και τι όχι. Ελπίζω να μην σας φανώ πολύ προκλητική, πολύ ε, προβοκατόρικες οι θέσεις μου. Αρχίζουμε μια θετική θέση ως εισαγωγή σχετικά με το ποια πράγματα λειτουργούν. Πρώτα, οφείλω να σας συγχαρώ, διότι χάρη στη σκληρή δουλειά σας η προστασία δεδομένων δέχεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή τις ημέρες αυτές. Βρίσκεται πραγματικά στο προσκήνιο των ε, πράξεων συμμόρφωσης πολλών επιχειρήσεων. Και αυτό είναι μέγα επίτευγμα, όπως ε, αντιλαμβάνεστε. Να σας πω λίγα λόγια σχετικά με την δική μου εταιρεία Schneider Electric. Είμαστε global leader σε αυτοματισμούς, δηλαδή είμαστε μεγάλη επιχείρηση και η πατρίδα μας είναι η Ευρώπη. Έχουμε γεννηθεί στη Γαλλία και επιχειρούμε σε, και στις 28 χώρες μέλη. Είμαστε όμως και παγκόσμια εταιρεία. Έχουμε 40.000 εργαζομένους στην επιχείρηση και 140.000 εργαζομένους στον υπόλοιπο κόσμο. Για μας η προστασία δεδομένων είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και την ε, παρακολουθούμε με μεγάλο ενθουσιασμό. Θα σας πω όσο γίνεται περισσότερες λεπτομέρειες στα επόμενα 8 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα σχετικά με την προσπάθεια συμμόρφωσης με τον κανονισμό και πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις χτίζουν την συμμόρφωση με την προστασία δεδομένων. Το πρόγραμμα προέρχεται από τα μέλη του Συμβουλίου μας και που ζήτησαν από το νομικό τμήμα να φτιάξουν ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις διατάξεις του GDPR. Οι επικεφαλής της εταιρεία, μεταξύ αυτών και εγώ, φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα με μια διευθύνουσα επιτροπή και με εκθέσεις προόδου και έχουμε μια ομάδα η οποία ασχολείται ειδικά με αυτό. Πώς οργανωνόμαστε λοιπόν. Βασικά έχουμε μια κεντρική ομάδα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας που έχει αναλάβει να σχεδιάσει το πρόγραμμα και δίνει την όθηση για το υπόλοιπο της εταιρείας. Δηλαδή γράφει, συντάσσει την πολιτική, συντάσσει τα template και συμβάλλει ώστε οι υπόλοιπε χώρε μέλη, δηλαδή η επιχείρηση τη υπόλοιπε χώρε μέλη και στον υπόλοιπο κόσμο, να εφαρμόσουν το πρόγραμμα και στις 28 χώρες μέλη, βέβαια έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που και εκεί επιχειρούμε, να φτιάξουμε ένα GDPR champion, πρωταθλητή GDPR και να είμαστε ηγέτες και στην, ε, στον χώρο του marketing, να προωθούμε δηλαδή τις κατευθύνσεις γραμμές που έχουμε συντάξει. Για να σας δώσω ε, κάποιους γονιδικούς αριθμούς, βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βεβαίως αυτό είναι αναλογικό με το μέγεθός μας έχουμε 300 άτομα τα οποία εργάζονται ειδικά για το πρόγραμμα συμμόρφωσης. Έχουν δηλαδή καθήκοντα ειδικά για να εφαρμόσουν τις ε, ε, σχετικές διατάξεις τις οποίες έχουμε εκπονήσει εμείς. Το πρόγραμμα μας συμμόρφωσης με τον κανονισμό βασίζεται σε ροές εργασίας work streams σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το κείμενο του GDPR. Να μην πω τώρα σε όλες τις λεπτομέρειες των workstream, αλλά για να σας δώσω κάποια ιδέα για το πώς λειτουργούν αυτά, το πρώτο workstream είναι βέβαια να φτιαχτεί ε, ένας οργανισμός που να έχει ως στόχο την ε, συμμόρφωση με τον ε, κανονισμό. Αλλά αυτό δεν είναι και το τέλος. Πρώτα-πρώτα έχουμε έναν GDPO, δηλαδή ε, αξιωματούχο, officer, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη συμμόρφωση σε όλες τις χώρες τις οποίες επιχειρούμε. Αυτά απαιτεί άλλωστε και ο κανονισμός. Έχουμε ένα δίκτυο ανταποκριτών προστασίας δεδομένων σε κάθε χώρα μέλος. Αυτή είναι σε διαρκή επαφή με τις επακεφαλείς και με τις αρχές προστασίας δεδομένων και διευθύνει όλους όσους ασχολούνται με τα θέματα αυτά σε κάθε χώρα. Μιλούν την τοπική γλώσσα και συνεννοούμεθα κάθε εβδομάδα μαζί τους για να διασφαλίζουμε ότι εκπληρούν αυτά τα καθήκοντά τους. Πάνω από αυτή την οργάνωση τώρα έχουμε και την λεγόμενη Privacy Committee, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των, της οργάνωσής μας και των μελών του Συμβουλίου που δίνουν τις κατευθύνσεις για όλους τους τομείς πολιτικής και για, όλους, για όλες τις statement για τους, για τους ε, πελάτες μας. Δεύτερο, επικοινωνία. Έχουμε ξεκινήσει μια μαζική επικοινωνιακή διαδικασία με όλους τους απασχολουμένους μας, ώστε να γνωρίζουν όλοι, όλοι τι σημαίνουν τα τέσσερα αυτά γράμματα. GDPR. Μέσω του διαδικτύου, μέσω ε, δικτύων που έχουμε οργανώσει εμείς για να μπορούν οι διάφοροι αυτοί να θέτουν ερωτήσεις σχετικά με το GDPR, να συγκεντρώνουμε τις απαντήσεις και να τις θέτουμε ως συχνά τιθέμενες ερωτήσεις, FAQs, για να μπορούν να τις παρακολουθούν και να παρακολουθούν και τις απαντήσεις. Έχουμε φτιάξει και ένα playbook για όσους εφαρμόζουν τις διατάξεις του GDPR για το πώς θα συντάσσουν τις ε, διάφορες ερωτήσεις, πώς θα συντάσσουν τις συμβάσεις με τους πελάτες και με τις άλλες επιχειρήσεις με τι οποίε συνεργαζόμαστε. Το χρονόμετρο βεβαίω προχωρεί αμήλικτα. Άλλο σημαντικό είναι η συμπλήρωση του Μητρώου, του Register, το οποίο καλούμεθα τώρα να ε, συντάσσουμε. Έχουμε φτιάξει λοιπόν τώρα τα σχετικά πλαίσια και ξεκινήσαμε από το λεγόμενο template, από το υπόδειγμα της γαλλικής αρχής. Θεωρήσαμε, εξετάσαμε μάλλον ποια πράγματα πρέπει να συμπληρώσουμε κάθε χώρα μέλο κάνει σχετικέ συμπληρώσει και λαμβάνουμε τακτικέ εκθέσει από όλε τι αρχές, από όλες τις, μάλλον, συγγνώμη, από χώρες τις οποίες δραστηριοποιούμεθα και κάνουμε τι σχετικέ συμπληρώσει και ζητούμε από τις ε, αντιπροσωπείε μα στις χώρε να ε, μα πούν αν χρειάζεται και τίποτε άλλο να συμπληρωθεί. Υπάρχουν βέβαια πολύ περισσότερα ε, στοιχεία του προγράμματος από αυτά που σας έχω αναπτύξει, δηλαδή φτιάχνουμε checklist, φτιάχνουμε πρότυπα, υποδείγματα. Έχουμε ε, δημιουργήσει και μια πολιτική για την ομάδα προστασίας δεδομένων, για την εφαρμογή του GDPR. Βεβαίως αυτή έχει και παγκόσμιο χαρακτήρα. Άλλο σημαντικό στοιχείο, άλλη σημαντική προσπάθεια που αναπτύσσουμε τώρα είναι η εξέβρεση μηχανισμών αυτοματοποίησης όλων αυτών, διότι βασιζόμαστε με το να βασίζεται κανείς σε αυτά τα υποδείγματα template δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό, τουλάχιστον από τη δική μας σκοπιά. Πολλές επιχειρήσεις αναζητούν προμηθευτές οι οποίοι να μπορούν να προσφέρουν εργαλεία, μηχανισμούς δηλαδή, που να μπορούν να, ε, να μας επιτρέψουν να βασιζόμαστε σε διάφορα, σε διάφορα εργαλεία ή αν μηχανισμούς αν θέλετε για την ε, εξέβρεση των δεδομένων και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί στην αγορά. Προσπαθούμε να τους βρούμε για να αναπτύξουμε κάποια από τα εργαλεία αυτά. Λίγα λεπτά μου μένουν ακόμη, θα προσπαθήσω να εξηγήσω ποια πράγματα τώρα δεν λειτουργούν. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, ο GDPR δεν τηρεί μια από τις δεσμεύσεις του μας υποσχέθηκε ένα ενιαίο πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ευρώπη, ώστε να διευκολυνθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να δραστηριοποιούνται δηλαδή στην ενιαία αγορά. Και δεν θεωρούμε ότι συμβαίνει αυτό. Θεωρούμε ότι είναι μάλλον το γαλλικό πρότυπο που το λένε «milfeuille» είναι αυτό δηλαδή που έχει πολλές διαστρωματώσεις, πολλά φύλλα αν θέλετε. Έχετε το ευρωπαϊκό, έχετε τα εθνικά επίπεδα χώρες μέλη με τις δυνατότητες ή την δυνατότητα προσαρμογής ε, ας πούμε του εθνικού ηλικίας, του εθνικού ορίου ηλικίας παιδιών, ανηλίκων κλπ. Αυτό όμως είναι δύσκολο γιατί είναι διαφορετικό αναχώρα μέλος και μας κάνει την ζωή πολύ δύσκολη. Μπορώ να σας τα αναπτύξω αυτά περισσότερο στο, στο στις ε, ερωτήσεις και απαντήσεις. Μετά υπάρχουν διάφορες εθνικές διαφορές πέραν του GDPR και γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο το σύστημα. Υπάρχει μετά και το άρθρο 29 και η ερμηνεία του GDPR. Μετά όλες οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων έχουν προχωρήσει σε ερμηνεία των εθνικών τους νόμων την οποία θέλουν να διατηρήσουν. Υπάρχουν μετά και οι εθνικές κατευθύνες γραμμές των εθνικών αρχών για τον GDPR, που καμιά φορά και αυτές έχουν μεταξύ τους διαφορές. Έχουμε το λευκό κατάλογο και τον μαύρο κατάλογο, που είναι όμως διαφορετικοί σε κάθε χώρα μέλος. Εγώ τώρα ως αξιωματούχος, ως GDPO που έχω αναλάβει την, ε, την συμμόρφωση με τον βασικό κανονισμό, πώς θα τα αντιμετωπίσω όλα αυτά. Όταν φτιάχνω μια πολιτική, χρειάζομαι καθαρούς, συνεκτικούς κανόνες βασισμένους στην Ευρωπαϊκή Συνένεση. Δεν μπορώ να έχω 28 διαφορετικέ πολιτικέ πρέπει να έχω μια πολιτική την οποία μπορώ να εφαρμόσω σε όλο μου το σύστημα ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων, IT, διότι ένα έχω μόνο. Ελπίζω να μας βοηθήσετε, εμάς δηλαδή τους αξιωματούχους προστασίας δεδομένων των επιχειρήσεων, να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε με τρόπο αποτελεσματικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ε, πολύ εμπεριστατωμένες και χρήσιμες παρεμβάσεις σας. Τώρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Θα οργανώσουμε τη συζήτηση με τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως. Όπως εξήγησα θα δίνω εναλλακτικά σε δύο εθνικούς βουλευτές και έναν ευρωβουλευτή μέχρι ότου εξαντληθεί ο κατάλογος των εγγεγραμμένων. Εάν θέλετε να λάβετε το λόγο ως μέλος Εθνικής Βουλής, σας παρακαλώ να δώσετε και πάλι το γαλάζιο έντυπο. Η κυρία Κοσοβόλη από την Ελλάδα. Ορίστε. Oh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, μιλήσαμε πριν ε, για την προετοιμασία και για την άμεση ε, εφαρμογή σε λίγες μέρες και καταδείχθηκε ότι πολλά πράγματα δεν έχουν γίνει ακόμη για την ενότητα με την οποία, για την οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να μεταφέρω ένα κλίμα από τη χώρα μου. Και αυτό έχει να κάνει με μία μελέτη που έγινε από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων σε επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες στην Ελλάδα το Φεβρουάριο ε, και θέλω να σας πω μερικά αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Είναι λοιπόν ενδεικτικό ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν γνωρίζει τον νέο κανονισμό ε, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 35% για επιχειρήσεις με λιγότερο από 100 εργαζόμενους. Ποσοστό 22% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τον ορισμό των προσωπικών δεδομένων και θεωρώ δε το ποσοστό που δηλώνει ότι γνωρίζει πρέπει να ελεγχθεί περισσότερο. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό, ενώ το 57,7% δηλώνει ότι συμμορφώνεται μερικώς. 8 στις 10 επιχειρήσεις αξιολογούν ως μέτριο ή χαμηλό το βαθμό ετοιμότητας ως προς τη συμμόρφωση. Αν συνυπολογίσουμε το κόστος συμμόρφωσης, που είναι περίπου 40.000 ευρώ, είναι προφανές ότι στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμη ώστε να επιτύχουν οι επιχειρήσεις τη συμμόρφωση αλλά και για να πιστούν για την αναγκαιότητά της. Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βγαίνουν από μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης και παρά τα σημάδια ανάκαμψης αντιμετωπίζουν ακόμα δύσκολες ε, οικονομικές συνθήκες. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις πρέπει να πιστούν ότι η εδραίωση μιας κουλτούρας σεβασμού και προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για αυτές. Ε, να αντιμετωπίσουν τον κανονισμό σαν ευκαιρία και σαν κίνητρο, ευκαιρία για επένδυση και δράσεις εκπαίδευσης προσωπικού και στα νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης απαιτείται ενημέρωση των υποκειμένων των δικαιωμάτων. Ε, εδώ θέλω να πω και άκουσα και προηγουμένως και μου προκαλεί εντύπωση ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση στις μεγάλες επιχειρήσεις από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις, για παράδειγμα ο ορισμός υπευθύνου στην μικρομεσαία επιχείρηση και αυτό το τονίζω γιατί στη χώρα μου ένα μεγάλο ποσοστό είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση που πριν ε, ε υπόθηκε νομίζω από τον κύριο ε, νομίζω ότι υπόθηκε από τον κύριο ε, Χέντριξ ε, ότι δεν υπάρχει στην πράξη αυτή η διαφοροποίηση. Νομίζω ότι και το άρθρο 29 και το 35 έχει σημαντικές διαφοροποίησεις. Ίσως στην πορεία επανεξετάσουμε τα δεδομένα αυτά, αλλά να μην πανικοβάλλουμε και να μην δημιουργούμε άγχος στις επιχειρήσεις αυτές. Θέλω λοιπόν, καταδεικνύεται από όλα αυτά και θέλω να το πω ότι ε, χρειάζεται μια καμπάνια ενημέρωσης. Δηλαδή η εποπτεύουσα αρχή κάθε χώρας, στη δική μας τη χώρα είναι αρχή προστασίας, η ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένων. Η ανεξάρτητη αρχή σε συνεργασία με τις επαγγελματικές ενώσεις των επιχειρήσεων πρέπει να κάνει μια μεγάλη καμπάνια επιμόρφωσης και πρέπει να διαμορφώσει και θεσμούς βοήθειας αυτών των επιχειρήσεων για μπορέσουν να εναρμονιστούν με τον κώδικα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Η, ε, η κυρία, ο κύριος Λαμπάρτα από την Ισπανία. Ορίστε, κύριος. Ομολογώ πως ε, με εκπλήσουν τα περιεχόμενα κάποιων εισηγήσεων που αναφέρθηκαν ε, στην πλήρωση των όρων ε, του κανονισμού σε σχέση με τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φαίνεται από ό,τι κατάλαβα ότι θα ε, εφαρμοστεί Πρόκειται για μια οδηγία η οποία εφαρμοζόταν εδώ και 33 χρόνια άμεσα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολλές από αυτές, περισσότερες από αυτές συντηρούσαν. Δεν υπάρχουν δεν υπάρχει κανένα νέο δικαίωμα το οποίο να ε, αυτός ο νέος κανονισμός σε σχέση με τον κανονισμό, την οδηγία που εφήρμοζαν αυτές οι εταιρείε ε, εδώ και 33 χρόνια. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, υπήρχε κάτι πριν. Δεν είναι λογικό λοιπόν να προκαλείται ένα τέτοιο ε, ε, πανικός ή ε, σε σχέση ας πούμε με αυτό το υποτιθέμενο φόρτο το γραφειοκρατικό γιατί ας πούμε η Ισπανική Αρχή έχει εισάγει στην πλατφόρμα της στην ψηφιακή ένα εργαλείο που ονομάζεται διευκόλυνση και που επιτρέπει στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείσουν ε, το θέμα σε 45 λεπτά σε σχέση δηλαδή με τις υποχρεώσεις η καινοτομία ποια είναι ότι πολλές από στις ε, καινούργιες χώρες ε, μπορεί να εφαρμόσουν ε, οικονομικές κυρώσεις. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία. Μπορούμε να το πούμε ως παιδαγωγική μέθοδος διατοσκύρωσης. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται. Ε, οι πιθανές κυρώσεις ενάντια μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι ελάχιστες με βάση τα όσα προβλέπει ε, ο νέος κανονισμός. Δεν είναι πάντα μόνο κυρώσεις οικονομικές, αλλά υπάρχουν και κυρώσεις άλλες φύσεις. Δεν νομίζω λοιπόν πως είναι ε, λογική αυτή η υπερβολική ε, ανησυχία. Γιατί μόνο σύγχυση προκαλεί. Είναι κανόνες που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν μπορούμε να ζητάμε εξαιρέσεις για κανένα τομέα. Κάτι τέτοιο δεν θα βοηθούσε σε, αυτή, σε, σε καμία περίπτωση. Δεύτερον, πιστεύω πως υπάρχει μια πτυχή, το αναφέρατε στην πρώτη παρέμβαση, που μας, ε, θα πρέπει να μας χαροποιήσει για το έναρξη ισχύω αυτού του κανονισμού, δηλαδή η ομοιομορφία των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Πώς θα γίνει με την οδηγία του 95 ε, υπήρχε ένας ε, ε, τροποποίηση μάλλον αυτής της οδηγίας θα υπάρξει ένας αντίκτυπος παγκόσμιο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Όμως θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια από πλευρά των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων αλλά και της Ευρωπαϊκής αρχή Δεδομένων ώστε να υπάρξει μια ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων και μη ευρωπαϊκές εταιρείε να ε, μπορέσουν να παίξουν το ρόλο τους και να ακολουθήσουν ε, και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του νέου κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα πάρει το λόγο η κυρία Κοράτζα Μπίλτ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και θα ήθελα να καλωσορίσω και μια ομάδα επισκεπτών που έχει προσκληθεί από την ίδια από την Σουηδία. Θα Σας καλωσορίζω λοιπόν ε, και σας. Ευχαριστώ πολύ Γιάννα Φίλιππ και για την εργασία που έχεις κάνει με την ε, ιστορική σημασία σε αυτή η νομοθεσία που θεσπίζει ε, ιστορικές προδιαγραφές τις ψηλότερες στον κόσμο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι προϋπόθεση για την ενιαία ψηφιακή αγορά και έτσι ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Εγώ είμαι μεταξύ όσων είναι πολύ ευχαριστημένοι για αυτόν τον κανονισμό. Έχουμε προσπαθήσει πολύ εδώ και στην Επιτροπή προστασία του Καταναλωτή για να μπορέσουμε να έχουμε όσο γίνεται πιο ισορροπημένο αποτέλεσμα. Δεν το καταφέραμε απολύτως να έχουμε βεβαιότητα νομική, να έχουμε μια ενιαία νομοθεσία και αυτός, γι' αυτό τον λόγο αλλάξαμε την προηγούμενη οδηγία και ε, ε, μετά από δύο χρόνια δεν έχουμε ακόμα μόνο τις μικρές επιχειρήσεις αλλά πούμε και ο Ερυθρός Σταυρός ε, σκέφτεται πώς θα κάνει και πώς θα προστατέψει τα στοιχεία. Οι σύνδεσμοι, οι σχολικοί δεν ξέρουν ο κόσμος τι να κάνει με τις κάρτες του. δεν τα ξενοδοχεία δεν ξέρουν τι να κάνουν με τους καταλόγους των επισκεπτών τους. θέλουν να κάνουν το σωστό αλλά αγωνίζονται, εξακολουθούν να αγωνίζονται. Οι μόνοι που κερδίζουν είναι οι διάφορες συμβουλευτικές εταιρείες. Είναι χρυσορυχείο για τους συμβούλους και δεν θα έπρεπε να, έτσι να ήταν τα πράγματα. Μια σουηδική εταιρεία μου είπε ότι δαπάνησε 5 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια οι Google και οι Facebook δεν έχουν πρόβλημα, αυτοί έχουν λεφτά με ουρά. Οι μικροί, οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που πρέπει να πληρώσουν την ύφη. Και αυτό είναι λάθος, γιατί εμείς άπρεπε έπρεπε να έχουμε ε, και να προσφέρουμε σαφήνεια στους συμπολίτες μας. Πρόκειται για έναν κανονισμό που βασίζεται σε εξαιρέσεις. Μόνο έτσι μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο. Επίσης ανησυχώ όσον αφορά την καινοτομία. Μια εταιρεία όπως η Spotify δεν, μπορούσε να, δεν θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί έτσι όπως αναπτύχθηκε αν είχε ισχύσει νωρίτερα το, ο κανονισμός τούτος. Ε, πιστεύω πως θα είναι λιγότερη αυστηρή η εφαρμογή, ότι θα υπάρχει μία εναρμονισμένη εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση, γιατί όπως υπόθηκε και πριν η εφαρμογή είναι πολύ κατακαιρματισμένη αυτή τη στιγμή. Αυτό Ελπίζω πως θα ισχύσει φιλική στάση και συμπεριφορά απέναντι στι εταιρείε που θέλουν να κάνουν το σωστό, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουν πώς θα το κάνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, διότι πρέπει να φύγει. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκίγια από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και μετά θα προχωρήσουμε στους υπόλοιπους εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, ε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας κάποιες παρατηρήσεις για την φύση αυτής εδώ της ε, ε, συνεδρίασης. Εμείς συγκαλέσαμε αυτή την διακοινοβουλευτική σύσκεψη με την ευκαιρία της συνθήκης της Λισαβόνας που άρχισε να ισχύει ακριβώς όχι για να μοιραστούμε γνώμες ή ανησυχίες αλλά και για να νεώσουμε τη δέσμευσή μας με την Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή ε, νομοθετική διαδικασία και την ίδια την ιδέα της ε, σύνταξης νομοθεσίας, της νομοθετικής διαδικασίας που σημαίνει ότι ε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτέλους θα εφαρμοστεί. Επιμένω για την ιδέα ε, της δέσμης, διότι πρόκειται για έναν κανονισμό και μία ε, οδηγία που απευθύνεται στις ε, υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου που είναι επιφορτισμένες με την διερεύνηση των αδικημάτων ή και ποινικών αδικημάτων. Το ε, πρώτο, το πρώτο σκέλος του πακέτου είναι κανονισμός και αυτό είναι διαφορά, είναι άμεσα εφαρμοστέος ο κανονισμός και οι πολίτες μπορεί να το γνωρίζουν ότι μπορεί απλά να προσφύγουν στο αρχικό σύστημα του κράτους μέλους ε, ώστε να εξασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Όμως, καθώς είναι κανονισμός, σημαίνει ότι κομμάτι της δουλειάς πρέπει να το κάνουν τα εθνικά κράτη-μέλη. Δεν, δεν, δεν αποκλείεται η εφαρμογή από τα εθνικά κράτη-μέλη ορισμένων μεταρρυθμίσεων που ε, υιοθετούνται με την έναρξη ισχύω του κανονισμού 25 Μαΐου. Δεύτερη ιδέα είναι πως ναι, πρόκειται για έναν κανονισμό που θα σημάνει τη διαφορά γιατί δεν απευθύνεται μόνο στις αρχές αλλά και στον ιδιωτικό τομέα συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό είναι σχεδόν ε, ηρωνικό γιατί όταν ε, υιοθετήσαμε αυτή τη νομοθεσία γνωρίζαμε ότι οι γίγαντες του ίντερνετ ήταν εναντίον μας. Ξέραμε τι σημαίνει να έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ισχυρή ε, αντίσταση του Google, της Amazon και των υπόλοιπων γιγάντων του ίντερνετ γνώριζαν τι συζητούσαμε εδώ και αυτό επηρεάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα δεν θα πρέπει να αγνοούμε τις δυσκολίες ε, ε, της επεξεργασίας ε, και του ελέγχου, ε, μάλλον τις δυσκολίες των ε, υπευθύνων επεξεργασίας στοιχείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ημερομηνία αυτή το 25η Μαΐου δεν θα πρέπει να τηρηθεί από όλους. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Έχουμε τονίσει από την Επιτροπή ότι θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να κατανοήσει αυτές τις δυσκολίες και τα προβλήματα όταν πρόκειται να επιβάλλει πρόστιμα. Χρειάζεται λοιπόν ε, ε, κατάρτιση ε, σχηματισμός δυνατοτήτων, η αύξηση της συνειδητοποίησης εξατίας και οι επενδύσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις σχετικές πολιτικές. Γιατί τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι, δεν είναι υποσυζήτηση. Υπάρχει ο χάρτης που είναι άμεσα, εφαρμοστέ, άμεσα εφαρμοστέος άρθρα 8 και 15. Ε, λοιπόν, αυτά δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Οπότε χρειάζονται επενδύσει από τα εμπορικά επιμελητήρια, χρειάζονται ε, επενδύσει από τις κυβερνήσεις και από ε, τα κοινοβούλια, δεσμεύσεις, έτσι ώστε αυτή η νομοθεσία επιτέλους να ταθεί σε εφαρμογή στη σωστή προθεσμία. 25 Μαΐου. Γι' αυτό είναι πολύ ουσιαδές να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εξασφαλίσουμε πως θα προστατευθούν σωστά τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με αυτόν τον νέο κανονισμό με την πλήρη συνεργασία και δέσμευση των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, the next speaker now... Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπούτινγκεκ από τη Μάλτα. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Πρώτα, να πω το εξής. Λαμβάνω τις αντιδράσεις των ε, μικρών επιχειρήσεων από τη χώρα μου, παρακολουθούν τη σημερινή συζήτηση και ένα ενδιαφέρον, ένας επιχειρηματίας μου λέει ότι ο GDPR χρησιμοποιείται για να εκφοβήσει ορισμένους και επειδή η παρατήρηση αυτή προέρχεται από μικρομεσαία επιχείρηση, θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να την ακούσουμε, διότι από τα μείζωνα σφάλματα που έχουμε κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο εθνικό επίπεδο είναι ότι δεν ακούμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Παρακολούθησα λοιπόν προηγουμένω τον κύριο Χέντριξ και νομίζω ότι αυτό το είπε, τα εργαλεία εντό εισαγωγικών στα οποία αναφερθήκατε πρέπει να διανεμηθούν, πρέπει να φτάσουν μέχρι το τελικό χρήστη. Οι μικρομεσαίοι δεν αντιλαμβάνονται πώς μπορούν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους. Είναι σημαντικό και πρέπει να μοιραστούμε και την θεμελιώδη αυτή παρατηρήση που κάνουν οι πολίτες. Δηλαδή οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Και σε όλους μας ζητούν στις ιστοσελίδες πατήστε το κουτάκι στο κουτάκι που λέει I agree, συμφωνώ, χωρίς να έχει διαβάσει κανείς όλα αυτά τα ψηλά γράμματα. Κανείς δεν το κάνει αυτό, κανείς δεν κάθεται να διαβάσει σε τι συμφωνεί. Μιλούμε εδώ λοιπόν για ανθρώπους οι οποίοι συμφωνούν, συγκατατίθενται σε πράγματα όπου δεν έχουν την παραμικρή ιδέα περί τίνος πρόκειται. Και δεν μιλώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες. Γνωρίζονται προσωπικά οι περισσότεροι μεταξύ τους και μπορούν να έχουν ή μπορούν να προσφέρουν και στον ε, τελικό χρήστη των υπηρεσιών τους προσωπικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει θέμα εκεί να εκμεταλλευτούν παράνομα τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό που χρειάζεται να μας αποσχολήσει είναι οι μεγαλύτερες και οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, με διαφορετικό τρόπο λοιπόν. Αυτό ίσως να βοηθήσει εν τέλει να προωθήσουμε με σωστό τρόπο την συμφόρφωση με τις διατάξεις του GDPR. Παρόλο που ο Ισπανός συναδελφός μας πριν είπε ναι, υπήρχαν βεβαίω, υπήρχε νομοθεσία και από πριν. Εδώ πρέπει να απαντήσω και ναι και όχι, διότι υπάρχουν αλλαγέ. Αν δεν υπήρχαν αλλαγέ, αν δεν είχαν επέλθει δηλαδή οι αλλαγέ, δεν θα προσαρμόζαμε τώρα εκ νέου την νομοθεσία μα. Έγιναν λοιπόν αλλαγέ. Και ίσω κάποιοι να ήταν οι ποιότεροι, αν λιγότερο. Αλλά η δική μου έκκληση είναι και ιδίω εξ ονόματο της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων τη χώρα μου που είναι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τις καλύτερες προθέσεις για να προσαρμοστούν στις διατάξεις του κανονισμού. Ας μην τους κάνουμε πιο δύσκολο το έργο τους, ας τις διευκολύνουμε. Προς Θεού, απλοποιήστε ολόκληρο το σύστημα. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Φόρε από ε, την Βελική Βουλή των Αντιπροσώπων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και πριν, βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας και η παρακολούθηση και αξιολόγηση θα έχουν μεγάλη σημασία για να δούμε με ποιον τρόπο εφαρμόζεται ο κανονισμός και βεβαίω η εταιρεία Schneider Electric που είναι παρούσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και εκτό Ευρώπης τα εξήγησε προηγουμένω. πώς δηλαδή μπορεί να προσαρμοστεί μια επιχείρηση με πιο εναρμονισμένο τρόπο στις ε, ανάγκες συμμόρφωσης του κανονισμού και θα πρέπει να βασιστούν και όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες στην ίδια προσπάθεια. ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στην νομοθεσία και στην ευρωπαϊκή επικράτεια σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ των εταιριών και από τη μεριά και των αρχών προστασίας δεδομένων από την άλλη. Για το ποιε θα είναι δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ εταιριών και αρχών και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, βεβαίω και μιλώ για μικρέ, μεσαίε και μεγάλε επιχειρήσει και εσεί βεβαίω, απευθύνομαι πάντοτε στην εκπρόσωπο τη Schneider Electric, θα, ε, εσεί θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε το πράγμα και παγκόσμια και γι' αυτό η πρώτη μου ερώτηση είναι για την νυν και τη μελλοντική σχέση σα με τι αρχέ προστασία δεδομένων. Μιλήσατε προηγουμένω και για κάποια ιδεώδη εργαλεία που θα έπρεπε να ε, ε αναπτυχθούν Έχετε κάποιες πρακτικές, κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από όλε τις ε, επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να μπορούν να βασιστούν και αυτές στην δική σας τεχνογνωσία. Τέλος, για την ψηφιακή κυριαρχία. Επιχειρήσεις ευρωπαϊκές όπως η δική σας, πώς θεωρείτε ότι θα ενισχυθεί αυτή η ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία από την εφαρμογή του, νέου, του, βασικού κανονισμού. Αυτέ είναι οι ερωτήσει που θα θέσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα, ο επόμενος, ή μάλλον η επομένη είναι η κυρία Στίβενς από την ομάδα ε, ε, ECR του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ομιλητές μας που ήρθανε δεν αρκεί να λέμε ότι ο κανονισμός ε, θα έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις μας. Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος ε, και ειδικά για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πριν από δύο εβδομάδες ο φλαμανδικός τύπος δημοσίευσε μια έρευνα για το πόσες επιχειρήσεις γνώριζαν το τι σημαίνει για την επιχείρησή του, ο νέο αυτός κανονισμός. Και το αποτέλεσμα ήταν πω μόνο μία στι τρει επιχειρήσει ε, ήξεραν το τι σημαίνει αυτό για την επιχείρησή τους. Είναι λοιπόν κάτι το πολύ σημαντικό, αλλά δεν επιτρέπεται να καταλήξει σε περιττή γραφειοκρατία για τις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και βεβαίω δεν είναι μόνο ε, η ευθύνη των κρατών μελών, αλλά και δική μας. Όλες οι αρμόδιες αρχές ε, θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν και να συμβουλεύσουν τις επιχειρήσεις ε, για να συνεισφέρουμε τελικά στην ε, λειτουργία τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πλούς και κατόπιν από την Πολωνία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε δέκα ημέρες πριν από την επίσημη εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού στην Ευρώπη και ακούγοντας την συζήτηση φοβούμε ότι θα αποτύχουμε ως Ευρώπη να έχουμε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων. Συμφωνώ με την κυρία Αναμαρία Κόρατσα Μπίλτ από την Σουηδία όσον αφορά την προετοιμασία και βεβαίως για το ότι μιλάμε για θησαυρό που θα κερδίσουν ε, τελικά οι εταιρείε ε, συμβούλων και θα καταλήξουμε σε μια τιμωρία των μικρών επιχειρήσεων. Ε, καταλήγουμε σε κάποιες γελίες καταστάσεις. Μου είπε η κόρη μου ότι το αξιολόγιο στο σχολείο πλέον θα είναι με αριθμούς, θα φωνάζουν αριθμούς και όχι όνομα. Ε, εντάξει κάποια στήριξη χρειάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή σας να ξεκαθαρίσουμε το τι σημαίνει αυτό για τις μικρές ε, εταιρείε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί όντως το πέρας να μην είναι τόσο μεγάλο όσο το περιγράφουν ε, ειδικά αυτοί οι οποίοι θέλουν να βγάλουν λεφτά από αυτή την υπόθεση με συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ε, προτείνω λοιπόν να γίνει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία, να εξηγήσουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε. Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δηλαδή προστασία των δεδομένων. Αυτό το χρωστάμε και στις επιχειρήσεις και στους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το αυτή η πανευρωπαϊκή εκστρατεία επεξήγηση, αν θέλετε θα πρέπει να είναι σαφής. Δεν θα έχουν τον χρόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διαβάσουν τα νομικά ή κανένα βιβλιαράκι. Πρέπει να είναι απλή και σαφής. Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Ενιών από την Γαλλία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πως αυτή η ανταλλαγή με τις εταιρείε είναι πολύ σημαντική για μας τους ε, βουλευτές που οφείλουμε να ε, τίνουμε βίκονους στις δυσκολίες εφαρμογής αυτού του κειμένου που είναι τόσο σημαντικό. Όμως ε, βρίσκω πως είναι κάπως προκλητικό το να συζητάμε σαν να είναι ένα κείμενο Google, το οποίο δεν ε, είναι καθόλου προσαρμοσμένο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν νομίζω πως η γκάφα, οι μεγάλες δηλαδή πλατφόρμες του ίντερνετ είναι τόσο ικανοποιημένες για αυτό το κείμενο ε, και θα επανέλθω σε αυτό που είπα στο πρώτο γύρο του τραπεζιού. Δηλαδή βάζουμε εδώ ως εκείμα το μέγεθος της εταιρεία, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να μετρήσουμε και το επίπεδο του κινδύνου που δεν είναι αναγκαστικά αντίστοιχο με το μέγεθος της εταιρείας γιατί υπάρχουν startup που θέλουν να ξεκινήσουν με εφαρμογές ε, για προφίλ ή για εκμετάλλευση των μεγάλων ε, δεδομένων, των big data που δεν ε, αποτελούνται παρά από 3-5 άτομα. Αλλά ο κίνδυνος της εφαρμογής είναι πολύ σημαντικός. Πιστεύω λοιπόν πως αυτή η ενημέρωση που πρέπει να γίνει προς τις εταιρείε που θα επιτρέψει την αποδραματοποίηση πραγματοποίηση αυτής της προσέγγισης που γίνεται από πολλούς συμβούλους που πιστεύουν ή ελπίζουν να εκμεταλλευτούν ε, την εφαρμογή αυτού του κειμένου, σίγουρα. Αυτό είναι ο ρόλος, ε, να τους κάνει να δουν ποιε ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, και να... Και είναι σημαντικό όλα αυτά να γίνουν καλά κατανοητά Έχουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε ακόμα πιστεύω στο θέμα της επικοινωνίας και να δώσουμε να γίνουν κατανοητές οι, οι στόχοι αυτού εδώ του κειμένου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι κλείνει ο κατάλογος των ομιλήτων. για, καθώς και ο χρόνος ερωταπαντήσεων. Θα σας δώσω το λόγο για να βγάλετε κάποια συμπεράσματα, αλλά αναφέρω πως βέβαια το μέγεθος μιας εταιρεία μόνο δεν μπορεί να είναι το κύριο θέμα, δεν φαίνεται να είναι το κύριο θέμα πια. Ίσως θα μπορούσατε να απαντήσετε να, να επιμείνετε μάλλον σε αυτό το σημείο ε, κάπως περισσότερο ε, και σας δίνω το λόγο με την ίδια σειρά. Ευχαριστώ. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας σε σχέση με τη με το, ε, σε σύνδεση με τις αρχές ελέγχου των δεδομένων, προστασίας των δεδομένων. Θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται πιο σφαιρική προσέγγιση και με σεβασμό στους υπαλλήλου, αλλά και στους παίκτες μας. Όπως σας είπα, αυτό ε, μπορεί να ισχύσει όχι μόνο εδώ στην Ευρώπη αλλά και παντού στον κόσμο και να έχουμε ως κατευθυντήριο μας ε, γραμμή της ε, προτάσεις της ΚΝΙΛ γιατί η έδρα της εταιρεία μας είναι στο Παρίσι. Άρα λοιπόν ε, ε εμείς υπακούμε στη γαλλική νομοθεσία. Δεν θέλουμε και γενικά πρέπει να αποφεύγουμε τη δημιουργία παραδείσων για τα προσωπικά δεδομένα έτσι ώστε χώρες και φορείς να μην μπορούν να καταφύγουν σε τέτοιες, ε, ή μάλλον οι εταιρείες να μην μπορούν να καταφύγουν σε χώρες όπου θεωρούνται παράδεση. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, να προστατευτούν οι οι ε, παίχτες μας και πρόκειται για πέντε δις ε, ε, παίχτες και δυνητικούς παίχτες πολύ σημαντικό να κατανοηθούν οι ανάγκες και το θέμα. Για μια ολόκληρη μέρα ήρθε η ΚΝΙΛ μάλιστα στην επιτερία μας και συζήτησε με τους ανθρώπους που είναι αρμόδιοι για αυτά τα θέματα. Στην αρχή υπήρξαν άνθρωποι που μας λένε τι γίνεται με τον έλεγχο, πώς θα γίνει με τον νέο κανονισμό. Υπήρξαν κάποιοι δισταγμοί και τελικά κατάλαβαν όλοι πως καλύτερο είναι να προσπαθήσουμε να συνοηθούμε. Εξηγήσαμε στους ρυθμιστές ποιε είναι οι ανάγκε μας και του θέσαμε και ερωτήσει για να δούμε πώς θα μπορούσαμε με το καλύτερο τρόπο να σεβαστούμε τα παιχνίδια αλλά και τον κανονισμό. Είναι περίπλοκη κατάσταση για κάποιους φορείς, όντως θα πρέπει να ε, δούμε και να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα. Πάντως από το 2004 που η Κνήλη είχε περισσότερα μέσα για επιβολή ε, κυρώσεων είδαμε ότι σέβονται πολύ καλά οι εταιρείε και μάλιστα τα πρόστιμα είναι όλα ένα και πιο ψηλά ε, ε, και κατά συνέπεια οι εταιρείε σέβονται και περισσότερο. Είναι κρίμα που αναγκάζονται να βάλουν πρόστιμα αλλά αυτό ενισχύει την ε, ε, προσέγγιση των ε, ε, ε, αρχών ελέγχου και την, ε, την προσαρμογή των εταιριών στους κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε οι φορείς οι οποίοι είναι εκτός της Ένωσης να λένε ότι εντάξει μας δεν μας νοιάζει γιατί εμείς δεν διεπόμαστε από αυτούς τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες γιατί μας η έδρα μας είναι εκτός Ευρώπης και ευτυχώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει λάβει διαφορετική θέση είπε ότι οι διάφοροι φορείς ακόμα και αν είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να σέβονται την οδηγία ε, και η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό πλονέκτημα γιατί ακριβώς όλοι μπορούμε να δουλέψουμε επίσης ώρες. Έπειτα ε, βέβαια η εφαρμογή ε, της κύρωσης, η επιβολή μάλλον της κύρωσης είναι διαφορετική υπόθεση αν κανείς είναι εκτός ένωσης. Αυτό που είναι περίπλοκο είναι να μπορούν να προτείνουν όλοι αυτοί οι φορείς να συνοδεύουν με επαρκή τρόπο τα όσα συμβαίνουν. Ε, πιστεύω δηλαδή πως οι εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων δεν έχουν αυτή τη στιγμή αρκετό προσωπικό για να μπορέσουν να ελέγξουν την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Χέντριξ, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν νομίζω πως υπευλήθη κάποια συγκεκριμένη ερώτηση προς εμένα, αλλά έγιναν πολλά σχόλια και θα ήθελα να απαντήσω. Τις ε, παρεμβάσεις ε, του συναδελφού από την Ισπανία μεταξύ άλλων. Είπα στην αρχή ότι εμείς ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις σεβόμαστε το κράτος δικαίου να είναι σαφές δηλαδή, πρέπει να συμμορφωθούν με την νομοθεσία οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Έχουμε την κριτική μας, αλλά ο κανονισμό υπάρχει, πρέπει να συμμορφωθούμε, ε, για να είναι σαφές. Ποτέ δεν ζητάμε και γενικώ και το ξέρουν όλε τις ε, Βρυξέλλε εξαιρέσει ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί δεν είμαστε η εξαίρεση, είμαστε ο κανόνας. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι νομοθεσία προσαρμοσμένη στο μέγεθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Η νομοθεσία αυτή δεν φτιάχτηκε για επιχειρήσεις μικρομεσαίου μεγέθους και συμφωνώ πλήρως με αυτό το οποίο ακούστηκε ήδη για τον γενικό κανονισμό και είναι κρίμα που δεν υπάρχει κάποιος εδώ από την Κομισιόν γιατί θα μπορούσαν να το επιβεβαιώσουν. Εμείς πάντα λέγαμε πως δεν πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις γιατί πράγματι εξαρτάται από τον κίνδυνο και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορεί να υπάρχει κίνδυνος. Να είναι σαφές αυτό. Το, μπορείτε να το δείτε αυτό και στο έγγραφο θέσεών μας. Αλλά όταν νομοθετούμε πρέπει να μπορούν όλοι να συμμορφώνονται. Τίποτα το καινούριο είπατε. Ε, με συγχωρείτε αλλά η κυρία Κοράτσα Μπίλντ είπε ότι επρόκειτο περί ε, ενός ιστορικού κανονισμού. Ε, κάποια άλλη ευρωβουλευτή είπε ότι εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το πράγμα εδώ και χρόνια. Μα αν δεν είναι τίποτα το καινούριο, τι κάνετε τόσο καιρό. Εάν δεν είναι κάτι το καινούριο, γιατί οι κατευθυντήριες γραμμές της ε, Επιτροπής του άρθρου 29 δεν είναι ακόμα έτοιμες. Γιατί δεν έκαναν μια αντιγραφή. Γιατί δεν είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να πούμε το εξής. Κοιτάξτε, τα βασικά κείμενα που να εξηγούν τον κανονισμό δεν είναι έτοιμα. Οπότε δεν μπορείτε να περιμένετε ε, από μία μικρή επιχείρηση να είναι έτοιμη τώρα. Δεν ζητάμε λοιπόν εξαιρέσεις, ζητάμε μόνο τους επόμενους μήνες οι επόπτες, οι εθνικοί, να συνεχίσουν να ενημερώνουν και να κάνουν συστάσεις. Όπως και σε άλλους τομείς πολιτικής. Δεν αρχίζουμε κατευθείαν να κόβουμε πρόστιμα. Όχι. Προσπαθούμε ως προσπαθούν οι επόπτες να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με την νομοθεσία. Αυτό ζητάμε. Γιατί θέλουμε ο κανονισμός αυτός να γίνει σεβαστός. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτείτε α, ότι δεν μπορούμε να είμαστε έτοιμοι χωρίς το κείμενο. Και η κυρία Στίβενς μίλησε για το 1 τρίτο των επιχειρήσεων ε, είναι έτοιμες. Ε, με τα δικά μας δεδομένα μόνο ένα 15% των επιχειρήσεων είναι έτοιμες και στην Ισπανία, ε, στην Καταλωνία λένε 25% μόλις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι έτοιμες και υπήρχαν εκστρατείες στην Καταλωνία ήδη. Πρέπει να αναγνωρίσετε ότι κάποια κείμενα δεν είναι ακόμα έτοιμα να ερμηνευτούν. Ε, και κάποιο φώναξε από κάτω να διαβάσουν την νομοθεσία. Ε, με συγχωρείτε, οι ε, επιχειρηματίε μα ήδη δουλεύουν 65 ώρε τη βδομάδα για να ε, μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους ε, καταναλωτέ του πελάτες και δίνουν και δουλειά, απασχόληση. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλουμε εμεί από του νομοθέτε είναι απλά κείμενα στην γλώσσα του. Αν δεν είναι έτοιμε, κάνει μεταφράσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκέλη, έχετε τον λόγο. Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευσή σας. Είχατε ένα κείμενο το 95 και δώσατε δύο χρόνια για τις εταιρείε και για τον δημόσιο τομέα για να εφαρμόσετε το κείμενο και ε, λέτε δεν είναι έτοιμο. Ρωτάτε λοιπόν γιατί. Ως ε, αντιπρόεδρος ε, της ε, Γαλλικής Ένωσης Εποπτών Προσωπικών Δεδομένων, να το εξής. ότι αυτό το οποίο παρατηρώ τα τελευταία 20 χρόνια είναι ότι υπάρχει μια καμπύλη θα έλεγα συμμόρφωσης ε, και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Επίσης υπάρχει μεγάλη αύξηση στους ε, διορισμούς και ορισμούς ε, υπευθύνων προσωπικών δεδομένων στις επιχειρήσεις. Στη Γαλλία, παραδείγματο χάρη, είχαμε πέρσι 2.600 μέλη, τώρα έχουμε 3.600 μέλη. Αυτό ε, δείχνει το ενδιαφέρον και πράγματι χρειάζονται επαγγελματίες για την προστασία των δεδομένων. Λοιπόν, γιατί οι εταιρείε και ο δημόσιο τομέα ε, δεν ε, ασχολούνται με το θέμα. Ναι, η οικονομία δεν πάει τόσο καλά. Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Υπάρχει επίσης έλλειψη γνώσης. Είναι κάτι το πολύ περίπλοκο. Προσπαθήστε να κάνετε μια ανάλυση προστασίας δεδομένων στην ιστοσελίδα σας. Δοκιμάστε το. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος και μπορεί να μην κάνετε και την σωστή ανάλυση. Συμφωνώ λοιπόν ε, με την ε, άποψή σας. Πράγματι, οι μικρομισές επιχειρήσεις και οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν δυσκολίες. Ε, δηλαδή, υπάρχει έλλειψη γνώσης. Ο φόβος του να μην γίνει κάτι λάθος, γιατί είναι και θέμα κρίσης το πώς ε, το κρίνει. Και ε, εντάξει, περιμένουμε κάποια κατεύθυνση. Γιατί αν δεν υπάρχει σωστή κατεύθυνση, κάνει κάποιος κάτι κατά και μπορεί να κάνει λάθος. Ε, δεν είναι λοιπόν πάντα εύκολο. Οπότε αυτός κάποια εξήγηση. Λοιπόν, να κατηγορήσουμε όλες τις εταιρείες που δεν κάνουν το σωστό ακόμα και όλους τους δημόσιους φορείς και τώρα έρχονται και λένε ξέρετε πώς θα συμμορφωθούμε. Κοιτάξτε, ε, είχα εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα πριν, ε, ήμουν εγώ ένας από αυτούς τους συμβούλους που λέμε και προτιμώ να έρθουν να μου πούνε πώς θα συμμορφωθούμε τώρα από το να κρύβονται και να μην συμμορφώνονται. Ε προτιμώ αυτήν την ε, προσέγγιση και να τους βοηθήσουμε να συμμορφωθούν στο μέλλον, ακόμα και αν έχουν καθυστερήσει χρόνια. Αυτή είναι η δική μου η προσέγγιση και ως επόπτης δεδομένων αυτή την προσέγγιση θα ακολουθήσω. Ρωτήσατε για το πώς θα διατηρηθεί η σχέση με τις αρχές προστασίας δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είμαστε κοντά στις αρχές ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρώτον, γιατί θέλουμε να αντιληφθούν τις ανησυχίες μας και να μοιραστούμε και τις ε, βέλτιστες πρακτικές μας και αντιστρόφως. Και βεβαίως οι μεγάλες εταιρείες ε, επί σειρά ετών ήταν ε, ο κινητήρας, ε, η κινητήρια δύναμη, για να φτιάξουμε κάποια υποδείγματα. Και βοηθάμε, ε, σημειώνεται πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. Και αυτό, όπως σας είπα, το βλέπω και ως πρόεδρος της Γαλλικής Ένωσης Εποπτών Προσωπικών Δεδομένων στις ε, εταιρείε. και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια αρχή η οποία θα αναλάβει τον ηγετικό ρόλο. Αυτό θα μας κάνει πολύ ευκολότερη τη ζωή μας. Ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η σχέση με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών. Οπότε υπάρχει μια βεβαιότητα εδώ για το εάν θα πρέπει να είμαστε σε επαφή μόνο με την γαλλική αρχή όπου είναι η έδρα της εταιρεία μας ή εάν ε, κάθε φορά που εισάγεται κάτι το καινούριο πρέπει να είμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ε, Και έχουμε ένα ερωτηματικό για τα εργαλεία, τα μέσα είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοια εργαλεία, ειδικά όταν δημιουργούμε μητρώα, ε, να μπορούμε να εργαζόμαστε σε πολλές γλώσσες. Παραδείγματος χάρη, ε, έχουμε ένα σύστημα πληροφορικής. Κατά κανόνα δεν είναι τοπικό. Οπότε πρέπει να μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με κάθε χώρα που χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα πληροφορικής σε πολλές γλώσσες, να συμπληρώνεται το μητρό και να μοιραζόμαστε όλες τις πληροφορίες με κάθε χώρα. Αυτό πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλες τις ε, γλώσσες. Εμείς χρησιμοποιούμε το εργαλείο ΚΝΕΛ για την αξιολόγηση αντικτύπου προστασίας δεδομένων. Ένα εργαλείο το οποίο γνωρίζω ότι πολλοί επίσης χρησιμοποιούν για να αναπτύξουν τα δικά τους, ε, τους δικούς τους μηχανισμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος ε, ζήτησε τον λόγο. Για ένα λεπτό όμως ε, μόνο για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να πω στον εκπρόσωπο των μικρομεσαίων πως που του φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπα. Ίσως δεν με κατάλαβε όμως γιατί. Εγώ έλεγα ότι ε, Ε, δεν είπα ότι δεν φέρνει τίποτα νέο ο κανονισμός. Είπα ότι για τις μικρομεσαίες στην ουσία δεν επιφέρει τίποτα το καινούριο. Γιατί από το 1978 οι μικρομεσαίες έπρεπε να τηρούν το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα ακύρωσης, ε, ένστασης, ε, την υποχρέωση να ενημερώνουν όταν ε, χρησιμοποιούν τα στοιχεία, εγγυημένα μέτρα ασφάλειας για τη διατήρηση του απορρίτου κτλ. κτλ. Αυτά υπήρχαν στην οδηγία. 23 χρόνια ιστορίας λοιπόν, από τα 95 με συγχωρείτε, πιστεύω πως αρχούν για να φτάσουμε σε έναν ε, κανονισμό. Το δικαίωμα στην λύθη ε, ήταν κάτι το οποίο περισσότερο ισχύει για την Google και όχι για τις μικρομεσαίες. Ε, γι' αυτό και δεν πιστεύω πως αυτός ο πανικός βοηθάει σε αυτή τη φάση. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ε, ήταν μια πολύ καλή συζήτηση. Αναφέρθηκαν πολλές ιδέες για το πώς θα γεφυρωθεί το κενό ανάμεσα στις μικρομεσές και τους ρυθμιστές αλλά και τους πολίτες. Ε, τέλος, να πω μόνο το εξής που αφορά τις κατευθύνες γραμμές και την ερμηνεία αυτών. Οι εξατίες ε, που αναφέρθηκαν και που ζητήθηκαν, φυσικά όλα αυτά μπορούν να γίνουν, αλλά όχι χωρίς χρήματα. Το να κατηγορεί κανείς τις εθνικές αρχές ε, ίσως να είναι εύκολο. Όχι, δεν κατηγορήσαμε. Ακούγεται μια φωνή, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πιστεύω καθήκον όλων μας ε, και ημών των αρμοδίων για τον ε, προϋπολογισμό να εξασφαλίσουμε ε, την ύπαρξη αυτών των πόρων. Μπορεί δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο και νομίζω πως είναι σημαντικό πόρισμα από τη σημερινή συζήτηση. Και φυσικά πιστεύω πως οι εθνικές αρχές ε, θα χρειαστεί να αποφασίσουν να μην επιβάλλουν κυρώσεις καταρχάς στις μικρο, μικρές εταιρείες που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να συμμορφωθούν, γιατί οτιδήποτε άλλο θα είναι δυσανάλογο. Πιστεύω λοιπόν πως οι εθνικές αρχές ε, αυτό ελέγχου θα το κάνουν αυτό και ότι θα μπορέσουμε ομαλά να εφαρμόσουμε τον κανονισμό στις 25 Μαΐου. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ, που συζητήσατε μαζί σας και τώρα στον τρίτο όροφο αυτού του κτηριού μπορείτε να πάρετε τα σανσέρ ή τις ε, σκάλες. Έχουμε ένα γεύμα που προσφέρεται στη διάρκεια του μεσημεριανού διαλύματος. Θα συνεχίσουμε στην, με τις απογευματινές συνεδρίες στις 2 ακριβώς σε αυτή εδώ την αίθουσα. Καλή σας όρεξη.